Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε που δεχθήκατε την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συζητήσετε μαζί μας, να συζητήσετε με τους Ευρωπαίους βουλευτές για την θέση της Ισπανίας στην Ευρώπη. Σήμερα είναι μια μέρα πολιτικά πάρα πολύ σημαντική, γιατί έχουμε πάντα ανοιχτό το θέμα του Brexit αλλά είναι σημαντικό για μας να μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουν σημασία, το θέμα της μετανάστευσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει και έχει ψηφίσει την μεταρρύθμιση του Δουβλίνου. Περιμένουμε τώρα τα, τις χώρες μέλη και το Συμβουλίο να υπερψηφίσουν και τη δική μας πρόταση έτσι ώστε να καταλήξει μια διαδικασία και μια συζήτηση γύρω από τα θέματα ε, των προσφύγων και της ε, μετακίνησής τους και της μετεγκατάστασής τους. Εμείς ζητάμε να περάσουμε από το 1,1 στο 1,3 του προϋπολογισμού για τους πόρους της Ένωσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα δημιουργήσει θέματα στα κράτη-μέλη, αλλά με τους ιδίους πόρους θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις διαφορές αυτές και εδώ η συζήτηση είναι πάντα ανοιχτή. Υπάρχει μια πρόταση λοιπόν από πλευρά του Κοινοβουλίου και αυτό που έχει σημασία για μας είναι να υπερασπιστούμε την θέση μας μια θέση κεντρική, μια θέση καρδιά της ευρωπαϊκής εξέλιξης Φυσικά έχουν περάσει τώρα και αρκετά χρόνια μετά από την ένταξη της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να χαιρετήσει και τον κύριο Μπορέλ, τον Υπουργό Εξωτερικών του Βασιλείου της Ισπανίας που ήταν πρόεδρος αυτήν εδώ την αίθουσα. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας εδώ και σας δίνω αμέσως το λόγο. Eh, κύριε Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, είναι τιμή, πραγματική τιμή η δυνατότητα που μου δίνετε να περθώ σε εσά για να σας μιλήσω για την ε, θέση της Ισπανίας σε αυτή την ε, συναρπαστική συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και είμαι πεπισμένος ότι είναι συναρπαστική και με βάση τη δική μου εμπειρία το 1985 όταν υπεγράφει η ένταξη Τη Ισπανία στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ήμουν 13 ετών. Και παρά το ότι πέρασε τόσο χρόνο, θυμάμαι πολύ σαφώ εκείνη τη μέρα. Θυμάμαι τη συγκίνηση που αισθανθήκαμε εμεί που κατά δεκαετίε ε, υποφέραμε λόγω έλλειψη τη δημοκρατία και των ελευθεριών στην Ισπανία. Θυμάμαι τη συγκίνηση μια γενιά, ε, ολόκληρη Ισπανών, τη γενιά των γονέων μου, ε, ανδρών και γυναικών, για του οποίου η Ευρώπη καθ' όλη τη διάρκεια τη δικτατορία σήμαινε ελευθερία, κράτος δικαίου, συνοχή και πρόοδος. Εκείνη τη στιγμή ε, εκπροσωπούσε πολλά για την Ισπανία. Ιδιαίτερα την εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει πισωγύρισμα. Ότι επιτέλους ήμασταν σε ειρήνη με την ιστορία μας. Ότι επιτέλους κανείς ποτέ δεν θα μας ε, αφαιρούσε τη δημοκρατία πλέον. Έκτοτε, οι επόμενες γενιές ε, Ισπανών, όπως η δική μου, είδαν τα εσωτερικά σύνορα να γίνονται ανάμνηση της ιστορίας και είδαν ε, να υπάρξει ότι υπάρχει αλληλεγγύη και σχέση με λαούς που παλιά ήταν μακρινοί. Πάντα ε, σε σεβασμό με τις αξίες που θεωρούμε ότι είναι σημαντικές, η νομική ε, ασφάλεια, ο διάλογος, η αποδοχή των άλλων, ο φεμινισμός, η ισότητα ευκαιριών, η αδελφότητα, η συνύπαρξη, η οικολογία και η αλληλεγγύη μεταξύ γενεών. Οπότε, βεβαίως, είμαι ένθερμος Ευρωπαίος. Είμαι περήφανος για τι εκπροσωπεί αυτό. Και ιδιαίτερα περήφανος τώρα που ορισμένοι προβάλλουν τον αντιευρωπαϊσμό για να επιτύχουν εκλογικά ωφέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε Ταγιάννη που μου δίνει την ευκαιρία να απευθυνθώ στο Κοινοβούλιο που είναι στην καρδιά αυτής της συζήτησης, που είναι μια μεγάλη πρόκληση. Τώρα που πρόκειται να εορτάσουμε την 40η επέτειο των πρώτων άμεσων ευρωπαϊκών εκλογών. Η Ένωση βασίζεται στην προτεραιότητα των δημοκρατικών αρχών. Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, πριν απ' όλα, θα ήθελα να αναφέρω την ψηφοφορία που έγινε χθε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Σέβομαι, αλλά σέβομαι ως ε, πρόεδρος της κυβέρνησης ενός κράτους μέλους, αλλά λυπάμαι επίσης για την ε, απόρριψη της συμφωνίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μια συμφωνία την οποία διαπραγματευθήκαμε για πάνω από 1,5 χρόνο. Και θέλω να αποδίσω φόρο τιμής στον ε, Μισελ Μπανιέ. Έκανε καταπληκτική εργασία για να διατηρήσει την ενότητα των 27 κρατών μελών. Όπως έλεγα, αυτή η συμφωνία ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευση για 1,5 χρόνο και νομίζω ότι είναι η καλύτερη εφικτή συμφωνία. Είναι η λύση που προστατεύει καλύτερα τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και του συνόλου των κρατών μελών τη Ένωση. Άρα τη Ευρωπαϊκή Κοινωνία. Είναι η λύση που προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών αλλά και τα δικαιώματα των ε, επιχειρήσεων. Είναι μια συμφωνία που έχει παραχωρήσει και από τι δύο πλευρέ. Είναι πολύ δύσκολο να επιτύχει κανεί κάτι τέτοιο, μια ισορροπία που επιδιώκει πρώτα απ' όλα μια συντεταγμένη έξοδο. Ε, άρα τώρα είναι θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου να εγκρίνει τι αποφάσει που θεωρεί κατάλληλε για τα επόμενα βήματα. Εμεί, ω κράτη-μέλη και ως ε, ενωσιακοί θεσμοί, κάνουμε τη δουλειά μα Και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνουμε τα αναγκαία μέτρα για να ελαχιστοποιήσουμε την επίπτωση μια ενδεχόμενη άτακτη αποχώρηση. Κυρίε και κύριοι, πάντα εξέφρασα τη γνώμη μου και στο Ισπανικό Κοινοβούλιο αλλά και στι διάφορε συνεντεύξει που έχω δώσει. Πάντοτε έχω τονίσει ότι είναι λάθο το Brexit και για την ε, Μεγάλη Βρετανία και για την Ένωση. Όλοι χάνουμε. Και ιδιαίτερα η Βρετανία όμω. Ιδιαίτερα εκείνοι που χρειάζονται περισσότερο την προστασία τη κυβέρνησή του. Δηλαδή οι πιο ευάλωτοι. Αλλά είναι μια κυρίαρχη απόφαση την οποία ε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να σεβαστούμε. Γι' αυτό επιθυμώ το Ηνωμένο Βασίλειο να διατηρήσει την πιο στενή σχέση με το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση όμω είναι δική του. Αλλά οι αρχέ μα είναι σαφεί. Η ε, ακαιρεότητα τη εσωτερική αγορά, ε, το αδιέρετο των τεσσάρων ελευθεριών και η αυτόνομη λήψη αποφάσεων από την Ένωση. Στα πλαίσια αυτών των τριών σημείων πάντα θα παραμείνουμε. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να σα μιλήσω για την ε, ανάγκη να κινητοποιηθεί η Ευρώπη. Για την ανάγκη να αποκτήσει νέα νομιμοποίηση η Ευρώπη ε, έναντι των νέων ε, προκλήσεων. Αλλά και έναντι εκείνων που θέλουν να καταστρέψουν την Ευρώπη. Υπάρχουν διάφοροι εντό και εκτό σημαντικοί παράγοντε που θέλουν να καταστραφεί η Ένωση. Ω επικεφαλή, ω συγγνώμη, ω ηγέτη τη σοσιαλδημοκρατική οικογένεια, Βεβαίω θα περιμένετε να μιλήσω για την κοινωνική Ευρώπη, για την Ευρώπη που προστατεύει και θα το κάνω γιατί η, Ευρώπη, η κοινωνική Ευρώπη είναι η Ευρώπη των πεπιθήσεων. Και γι' αυτόν τον λόγο, για αυτή την ε, ηθική ε, πεποίθηση, γιατί θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη αυτό που αναμένουν οι πολίτε ε, από αυτήν, διαρωτάμε ποια είναι η κεντρική ιδέα τη ομιλία μου. Θα είναι κάτι πολύ πιο απλό. Το συνοψίζω σε μια φρόση. Η Ευρώπη, για να μπορεί η Ευρώπη να προστατεύει, σε αυτή την ιστορική συγκυρία πρέπει εμεί να προστατεύσουμε την Ευρώπη. Πρέπει δηλαδή να φτιάξουμε μια Ευρώπη δικαιωμάτων που να προστατεύει του πιο ευάλωτου να προωθήσουμε μια Ευρώπη που να δίνει ευκαιρίες για τους νέους μας και για τους ε, μακροχρόνια άνεργους. Σε χώρε όπως η δική μου, οι μακροχρόνια άνεργοι δεν είναι μόνο 60 ετών, μπορεί να είναι και 45 και ε, πάσχουν από την Ευρώπη. Πρέπει να έχουμε μια κοινωνική Ευρώπη που να ενισχύει τον κοινωνικό ιστό αλλά και τον ε, ε, επιχειρηματικό ιστό και να προστατεύει εκείνους που πάσχουν από την επισφάλεια. Πρέπει να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την ε, άμυνα των συμπολιτών μας, ούτω ώστε η Ευρώπη να γίνει ένας ε, παγκόσμιος παράγοντας που να μπορεί να σεβαστεί τις αξίες και τα ιδανικά του. Η προστασία της Ευρώπης είναι να τονίσουμε ότι πιστεύουμε στη Συμφωνία των Παρισίων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και πρέπει να ολοκληρώσουμε μια για πάντα την οικονομική και νομισματική ένωση. Μόνο έτσι, με μια Ευρώπη που να ε, με τους πολίτες της, μια αυτόνομη Ευρώπη που να υπερασπίζεται το κοινωνικό του μοντέλο, μια Ευρώπη που θα ολοκληρώσει την οικονομική και νομισματική τη ε, δομή, μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει που θα έχουμε την ε, επόμενη δεκαετία με επαρκή εγγύηση. Τι επόμενε δεκαετίε. Δεν πρέπει λοιπόν να αμφιβάλλουμε. Στου εχθρού τη Ευρώπη, πρέπει να του πω, η πεποίθησή μα και η αποφασιστικότητά μα θα νικήσουν την, ε, τον αυταρχισμό. Ορισμένοι έχουν μια ρητορική που αποκλείει άλλου. Ορισμένοι έχουν ε, πολλοί συζητήσιμε μεθόδου και λένε ψέματα. Είναι η στιγμή εμεί να αποδείξουμε την πεποίθησή μα, την αποφασιστικότητά μα για να υπερασπίσουμε το κοινό μα εγχείρημα που είναι η Ευρώπη. Σήμερα γίνεται μια πραγματική μάχη ε, ιδεών. Αυτό είναι ένα πλαίσιο ε, που έχουμε σε όλε μα τι χώρε και σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Ε, πρέπει να υπάρξει οπισθοχώρηση ή πρόοδο. Εμεί θέλουμε το, να είναι σαφέ ότι το μέλλον ποτέ δεν κατακτήθηκε με υποχωρήσει. Γι' αυτό δεν θα κάνουμε καμία υποχώρηση στην ε, υποστήριξη του ευρωπαϊκού μοντέλου. Η Ευρώπη προστατεύει του πάντε. Όλοι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό, όχι μόνο τα κράτη-μέλη, όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια, όχι μόνο η κοινωνία των πολιτών. Το σύνολο τη κοινωνία πρέπει να προστατεύσει την Ευρώπη. Σε αυτού που στέλνουν μηνύματα εσωστρέφεια, ε, ακόμη και από εδώ, η Ευρώπη για μένα δεν είναι ούτε ποτέ θα είναι απειλή στην καταπληκτική πολυμορφία των χωρών μας, των γλωσσών μας και των πολιτισμών μας. Η Ευρώπη είναι ακριβώς το αντίθετο. Η Ευρώπη ε, αυξάνει, πολλαπλασιάζει, δεν διαιρεί τις ταυτότητες. Αν είσαι Ευρωπαίος δεν είσαι λιγότερο Ισπανός, το αντίθετο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν ήταν και δεν θα είναι απλώς μια γεωγραφική έκφραση. Ήταν και είναι κοινότητα αξιών. Των αξιών της ε, Γαλλικής ε, Επανάστασης, ελευθερία, ισότητα και η αδερφότητα που είναι τόσο σημαντική σήμερα. Αυτέ είναι οι αξίε ανοιχτών κοινωνιών, αισιοδόξων κοινωνιών που καινοτομούν, που δημιουργούν, που θεωρούν ότι το μέλλον είναι ευκαιρία, ποτέ απειλή. Είναι κοινωνίε που συνδέουν την αναγκαία ανταγωνιστικότητα για την οικονομική ανάπτυξη με κάτι που είναι θεμελιώδε, που μα καθορίζει ω Ευρωπαίου, που είναι η κοινωνική συνοχή και το μοντέλο μα ευημερία. Αυτή η δέσμευσή μα που μα ενώνει Όπω για παράδειγμα οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη ε, του θεματολογίου 2030, που είναι ένα πραγματικό συμβόλαιο τη ε, επόμενη δεκαετία που θα κάνει την Ευρώπη τον κύριο ε, πρωταγωνιστή αυτή τη προσπάθεια. Είναι προφανέ ότι υπάρχει κοινωνική απογοητεύση στα πλαίσια τη παγκοσμιοποίηση. Το βλέπουμε στι πόλει μα, στου δρόμου μα, στι πλατείε μα. Αυτή η απογοήτευση ευνοεί βεβαίω τη ρητορική των ακραίων έχουμε μια τεράστια, ένα τεράστιο παράδοξο. Πρώτα απ' όλα η παγκοσμιοποίηση ανακατένει με την, τον πλούτο μεταξύ περιοχών του κόσμου, άρα μείωσε την παγκόσμια ανισότητα, αλλά αυξάνει την ανισότητα, αυξάνει συγγνώμη, την, την ανισότητα στο εσωτερικό των κοινωνιών μα. Και αν το σκεφτούμε καλά, η αύξηση του αντιευρωπαϊσμού οφείλει πολλά σε αυτό το τελευταίο φαινόμενο. Αλλά η παγκοσμιοποίηση δεν είναι θεομηνία που μας βρίσκει ανυπεράσπιστους. Ο Γκέτα έλεγε ότι τα... οι γονεί θα πρέπει να δουν στα παιδιά του ρίζε και φτερά. Παρόμοια, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει στου πολίτε τη ρίζε, δηλαδή μια βάση στήριξη, μια προστασία, αλλά και φτερά. Δηλαδή να τους δώσει δυνατότητε για να, είναι, ε, ε, να έχουν ευμάρεια και να έχουν δυνατότητες σε έναν παγκοσμιμένο... Ε, είμαστε σε μια κοσμοϊστορική αλλαγή. Στι 26 Μαου θα ανοίξει ένα νέο κύκλο πολιτικό για την Ευρώπη. Και θα πρέπει να ελέγξουμε λοιπόν την παγκοσμιοποίηση για να εξακολουθήσει να ισχύει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Θα πρέπει να εδρεώσουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση συμπληρώνοντά την με την αναγκαία πολιτική, κοινωνική και θα ήθελα να προσθέσω περιβαλλοντική ένωση. Μία δεκαετία μετά την αρχή τη. πολλοί από του συμπολίτε μα εξακολουθούν να ε, υποφέρουν από τις επιπτώσεις της κρίσης λόγω ε, ανισότητας στους μισθούς, ε, μείωσης των μισθών και επισφάλειας. Η κρίση αυτή συνέδεσε την Ευρώπη με την ιδέα της ε, λιτότητας. Βεβαίως, ορισμένοι πάντα αντιμετώπιζαν λιτότητα γιατί ήταν φτωχοί. Αντιμετώπισαν όμω και αυτού οι οποίοι ποτέ δεν, ήταν, δεν αντιμετώπιζαν λιτότητα και ήταν υπεύθυνοι για την χρηματοπιστωτική κρίση που έθιξε όλε μα τι κοινωνίε. Το αποτέλεσμα ήταν, ήταν η ανισότητα. Ιδιαίτερα η ανισότητα μεταξύ γενεών, δηλαδή η ανισότητα των νέων, δηλαδή επιπλέον η ανισότητα των φίλων. Γιατί οι γυναίκες θίγονται πολύ περισσότερο, πολύ πιο έντονα από την ε, επισφάλεια και την ε, ανισότητα στην ε, ευημερία. Και γι' αυτό το λόγο υπήρξαν ε, διαιρέσει ε, στι κοινωνίε μα και μα διαίρεσε και εμά. Διαίρεσε τι χώρε του Νότου και τι χώρε του Βορρά, τη Ανατολή και τη βύση, του δανειστέ από του δανειζόμενου. Άρα πρέπει να κλείσουμε αυτή την φάση. Πρέπει να αποκτήσει νέα νομοποίηση Ευρώπη μεταξύ των πολιτών τη. Για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να απαιτήσουμε μια κοινωνική Ευρώπη, μια Ευρώπη των δικαιωμάτων. Η κοινωνική και εδαφική συνοχή είναι ουσιώδη πυλώνα. και είναι νομίζω παράδειγμα μοναδικό στον κόσμο τον, ότι οι ευρωπαϊκέ κοινωνίε έχουν τέτοια συνοχή. Πρέπει να υπάρξει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Δηλαδή, η παγκοσμιοποίηση με την ευρωπαϊκή προστασία να είναι ευκαιρία και όχι απειλή. Πρέπει να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή με σαφεί στόχου, μετρήσιμου για την απασχόληση, την κοινωνική δικαιοσύνη και για την βιωσιμότητα του κράτους κοινωνικής προνοίας. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε αυτήν την ε, πλευρά στις ευρωπαϊκές οικονομικές πολιτικές και στην πολιτική συνοχή. Αυτή είναι η φιλοσοφία της πρότασης που ε, πρότεινε στο Συμβούλιο η Ισπανική Κυβέρνηση η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού επιδόματος ανεργίας, ένα πραγματικό backstop για τους συμπολίτε μας, ούτως ώστε να αποκτήσει περιεχόμενο η τόσο σημαντική έννοια της αλληλεγγύης και της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Είναι μια ιδέα που θα προτείνουμε παράλληλα με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να ολοκληρώσουμε το καθήκον που μας ανέθεσαν τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα, την οδηγία συνδυασμού της προσωπικής και εργασιακής ζωής και την οδηγία για διαφανείς και προβλέψιμες ε, συνθήκες εργασίας. Πρέπει να διαβεβαιωθούμε ότι όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από τη φυλή τους, το φίλο τους και την ηλικία τους, θα πρέπει να έχουν ε, αξιοπρεπή εργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταπολεμήσει την επισφάλεια στην εργασία, την ε, ανασφάλεια, γιατί δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να κυριαρχήσει η ιδέα ότι οι νέοι θα ζήσουν χειρότερα από τι προηγούμενε γενιέ. Είναι θεμελιώδε και αυτή είναι η θέση τη Ισπανική κυβέρνηση. Να, να προωθηθεί η εγγύηση για του νέου. Κυρίε και κύριοι, πριν από 7 μήνες η Ισπανία απέκτησε μια κυβέρνηση με τις περισσότερες γυναίκες από όλες τις ε, κυβερνήσεις των χωρών όσα είναι ένα ορόσημο σε μια πορεία που έχει ακόμη πολλά βήματα μπροστά της. Ποτέ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την πορεία εάν δεν είχε δώσει την ιδέα και την έμπνευση η Ευρώπη. Σήμερα εδώ μέσα θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την προσπάθεια που κάνουν οι γυναίκες βουλευτές όλης της Υπήρου ούτω ώστε να προωθηθεί ο ε, φεμινισμός που είναι μέρος του κοινωνικού κεκτημένου. Σήμερα σας διαβεβαιώ ότι η Ευρώπη δεν θα κάνει κανένα βήμα πίσω. Θα κάνει περισσότερα βήματα μπροστά. Χρειαζόμαστε βοήθεια της Ευρώπης. Γι' αυτό σήμερα προτείνω να εγκρίνουμε μια στρατηγική ισότητας φίλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δεσμευτικό χαρακτήρα. Μια στρατηγική για να καταπολεμήσουμε το χάσμα μεταξύ των γενεών και την ε, μεγαλύτερη απασχόληση και επισφάλεια ε, που επηρεάζουν ιδιαίτερα τις γυναίκες. Η φωνή της Ευρώπης να είναι επικεφαλής στον αγώνα για το να γίνει 21ος αιώνας αιώνας των γυναικών. Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικέ οι αρχέ του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ισότητα ευκαιριών για την πρόσβαση στην αγορά εργασία και σωστέ συνθήκε εργασία και η προστασία και η κοινωνική συμπερίληψη των πάντων. Επαναλαμβάνω, γι' αυτό βασίζομαι στον κανονισμό τη Ευρωπαϊκή Αρχής ε, για την Εργασία για να εγγυηθούμε τα δικαιώματα των εργαζομένων στον αγορά εργασία. Η Ευρώπη θα πρέπει να ξέρει να δώσει περισσότερε ίσε ευκαιρίε και να τι εγγυάται στην πρόσβαση σε όλε τι μορφέ μόρφωση, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου, στον πολιτισμό, στην ε, επιστήμη, στην έρευνα συμφωνούμε όλοι ότι έχουμε ένα προπύργιο ουσιώδες έναντι εκείνων που θέλουν να καταστρέψουν το ευρωπαϊκό όνειρο. Κυρίες και κύριοι, για να δώσουμε εγγυήσει για την ασφάλεια των πολιτών μας και να ενισχύσουμε το ρόλο μας στον κόσμο, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα στην Ευρώπη της ασφάλειας και στην Ευρώπη της άμυνας. Εδώ και ένα χρόνο Ξεκινήσαμε την μόνιμη διαφθορτική συνεργασία για να δημιουργήσουμε ικανότητες στον τομέα της άμυνας μετά από δεκαετίες παράλυσης. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε αποφάσεις τώρα να προχωρήσουμε ξεκάθαρα στη δημιουργία ενός πραγματικού ευρωπαϊκού στρατού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δείξει στον κόσμο ότι είναι μια soft power εξ επιλογής και όχι εξ αδυναμίας. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το ρόλο μας και πέραν των συνόρων μας και η πολιτική βούληση για να το πετύχουμε αυτό είναι προϋπόθεση για την ενίσχυση του ρόλου μας διεθνώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ελκυστικό πρότυπο για τον κόσμο σε πάρα πολλά επίπεδα. Είναι ακριβώς η Ένωση που θα μας επιτρέψει να έχουμε ένα ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή εκπροσωπούμε τις δυνατότητες που παρέχει η πολυμερής συνεργασία και η πολυμερής διεθνής τάξη που βασίζεται στο δίκαιο και στους ε, κοινά αποδεκτούς κανόνες. Η Ισπανία, πρέπει να το πω αυτό, θα συνεισφέρει προς την κατεύθυνση αυτή για την ενίσχυση του ηγετικού ρόλου λόγω και των ε, <clears throat> ειδικών σχέσεων που έχουμε με τη Λατινική Αμερική, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις και το βάρος της Ευρώπης είναι πολύ κατώτερο από αυτό που θα της άξιζε. Και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε να είμαστε ένας πραγματικός παγκόσμιος εταίρος. Για να το πετύχουμε πρέπει να καταργήσουμε τον κανόνα της ομοφωνίας, όχι μόνο στην εξωτερική πολιτική, αλλά και σε θέματα φορολογίας, σε θέματα πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού, και στα θέματα του ελέγχου του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να προστατεύσουμε την Ευρώπη λοιπόν και να της δώσουμε διαδικασίες λήψης αποφάσεων ευέλικτες έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία, τη νέα αυτή κυριαρχία. Τρίτον, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την αρχιτεκτονική του ενημέου νομίσματος και να προχωρήσουμε στα πλαίσια του πολιετούς οικονομικού προγραμματισμού εδώ και 50 χρόνια στην Χάγη οι εκπρόσωποι της δικαστικής εξουσίας των κρατών μελών και των κυβερνήσεων της οικονομικής τότε Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησαν τη διαδικασία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Και από τότε κάθε δεκαετία, στο τέλος κάθε δεκαετίας υπάρχει ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Το 69 η κορυφή της Χάγης, το 79 το ενιαίο νομισματικό σύστημα, το 89 το σχέδιο Ντελόρ και το 99 η ίδρυση επίσημα του ευρώ. Βέβαια το κενό του 2009 δείχνει ακριβώς ε, τα προβλήματα τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν όταν η διεθνής δημοσιονομική κρίση απέδειξε και έφερε στην επικαιρότητα τις αδυναμίες της αρχιτεκτονικής ε, του ευρώ. Έτσι μπορούμε να δούμε καλύτερα τις επιπτώσεις της κρίσης ε, λόγω ακριβώς αυτής της ε, έλλειψης θετικού συμβάντος το 2009. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε λοιπόν το 2019 ε, και πρέπει να πούμε ταυτόχρονα ότι το ευρώ είναι μια επιτυχημένη προσπάθεια που ωφελεί οικονομικά και πολιτικά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις γιατί αλλιώς θα μείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ατελής <clears throat> και εκτεθειμένη ε, στην αστάθη. Το θέμα δεν είναι να ενισχύσουμε μόνο το δημοσιονομικό σύστημα, αλλά να μπορέσουμε μέσω της Τραπεζικής Ένωσης να προχωρήσουμε <clears throat> στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων εφόσον υπάρξουν κρίσεις στο μέλλον. Ε, νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε η Ευρώπη να ανακτήσει το ρόλο της σε αυτόν τον τομέα και οι πολίτες θα πρέπει να είναι ε, γνώστες αυτών, πρωταγωνιστές αυτών των μεταρρυθμίσεων που θα προστατεύσει τις καταθέσεις τους, θα τους προστατεύσει από τον πληθωρισμό και από τις ε, κειμενόμενες οικονομικές κρίσεις. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις. Η μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης θα βοηθήσει και να προχωρήσουμε σε επίπεδο καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτή είναι η σωστή στιγμή όταν έχουμε συγκεκριμένες ευνοϊκές οικονομικές προϋποθέσεις. Θα πρέπει να προλαμβάνουμε τις οικονομικές αλλαγές θα πρέπει να συμπληρώσουμε τη δομή του ευρώ πριν από την επόμενη κρίση η οποία μπορεί να αποδυναμώσει το νόμισμά μας και την ένωσή μας. Μαθαίνουμε από τις εμπειρίες που είχαμε μέχρι τώρα και προχωράμε με αποφασιστικότητα. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδρανείς. Αυτό είναι απαραίτητο και για τα ευρωπαϊκά όργανα αλλά κυρίως για τους αυτούς τους οποίους εκπροσωπούμε τους ίδιους τους πολίτες. Σχετικά με το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο νομίζω ότι έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας. Θα πρέπει να ενισχύσουμε στρατηγικές πολιτικές όπως η κοινή αγροτική πολιτική και οι πολιτικές συνοχής πολύ σημαντικές για χώρες όπως η Ισπανία. Οι αστικές περιοχές δεν θα πρέπει να απομακρυνθούν από την Ευρώπη της υπαίθρου. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι αν μειώσουμε τον προϋπολογισμό θα δεχθούμε μια Ευρώπη της οποίας θα μειούται συνεχώς η σημασία. Αυτό δεν πρέπει να σταλεί σαν μήνυμα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ικανοποιεί την Ισπανική κυβέρνηση γιατί έχει καλά στοιχεία όπως η εξωτερική πολιτική, η μεταναστευτική πολιτική, το επίπεδο των δαπανών, η ενίσχυση κάποιων προγραμμάτων καινοτομίας και η τεχνολογική ανάπτυξη. Πρέπει η Ευρώπη φυσικά να είναι κυρίαρχη στον τομέα της καινοτομίας και να μειώσει την εξάρτησή της στον τομέα της ε, ψηφιακής οικονομίας, ε, ε, της κβαντικής πληροφορικής και της κυβερνοασφάλειας και του αυτοματισμού. Μόνο όταν προχωρήσουμε τότε θα υποστηρίξουμε σωστά και τις προτάσεις για, την διπλασια... για τον διπλασιασμό του προγράμματος Εράσμους. Υπάρχουν φαινόμενα λοιπόν τα οποία οδηγούν δυστυχώς στην αύξηση της ανισότητας και στην παιδική ένδια. Νομίζω ότι η Ευρώπη των ευκαιριών, η πραγματικά καλή για τους πολίτες Ευρώπη ξεκινάει από την παιδική ηλικία. Και γι' αυτό ακριβώς η εγγύηση για την παιδική ηλικία είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει την καταπολέμηση του αποκλεισμού, του κοινωνικού αποκλεισμού. Κυρίες και κύριοι, η πρόταση την οποία έχουμε μπροστά μας έχει κάποια κενά, αλλά είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης και πρέπει όμως να υπάρξει ένα άλμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αξίζει πολύ περισσότερο από το 1% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Πρέπει να είμαστε σωστοί στις δαπάνες, πρέπει να ικανοποιήσουμε όμως και τις προτεραιότητες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από τα δίκτυα τα οποία έχουμε δημιουργήσει. Θέλουμε έναν προϋπολογισμό λογικό, προληπτικό, ο οποίος να δημιουργεί ευκαιρίες, να δημιουργεί συνέργειες και εξοικονομήσεις κλίμακας. Έτσι θα προχωρήσουμε στην προστασία της Ευρώπης, μια Ευρώπη κοινωνική, μια Ευρώπη άμυνας, μια Ευρώπη οικονομική και νομισματική. Θα πρέπει εμείς να έχουμε ένα σωστό επίπεδο ανάμεσα στα μέσα και στους στόχους. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να επανέλθω στην ιδέα να αντιμετω... για, το για το τελευταίο κομμάτι της παρέμβασής μου σε σχέση με θέματα όπως οι προκλήσεις στις κλιματικές αλλαγές και στη μετανάστευση. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να βασιστούμε στις ευρωπαϊκές αρχές. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα ιδεολογικά σύνορα. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνίες και σε συνενέσεις που ε, θα ξεπεράσουν τις διαιρέσεις. Βέβαια οι τομεί αυτή είναι το πεδίο μάχης για αυτούς οι οποίοι δεν πιστεύουν και δεν θα πιστέψουν ποτέ στην Ευρώπη. Είναι το χαρακτηριστικό αν θέλετε κομμάτι αυτών που θέλουν να υπονομεύσουν την φιλελεύθερη δημοκρατία. Και για μια ακόμη φορά το σημαντικό είναι να προστατεύσουμε την Ευρώπη, να προστατεύσουμε το ευρωπαϊκό πρότυπο και τις ευρωπαϊκές αξίες. Στον τομέα των κλιματολογικών αλλαγών στα διεθνή φόρα ακούγονται όλο και περισσότερο κάποιες θέσεις σκεπτικιστικές για να μην πω ξεκάθαρα πολεμικές. Η προοπτική μας στο πλαίσιο αυτό είναι να οδηγηθούμε σε μια συμβιβαστική πρόταση που να ανοίγει ευκαιρίες για το μέλλον. Η ενεργειακή μετάβαση είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για τον εξυγχρονισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και της δικής μας χώρας, τα ενεργειακά δίκτυα και οι διασυνδέσει θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα της χρήσης της ενέργειας και θα μειώσουν τις εκπομπές. Νομίζω ότι οι συνέπειες αυτών των προκλήσεων αν δεν αντιμετωπιστούν θα είναι καταστροφικές. Νομίζω ότι θα πρέπει και σε επίπεδο πολιτικής ένωσης να πάρουμε μέτρα έτσι ώστε ο αυταρχισμός και ο υπερβολικός εθνικισμός που αποκλείει από την ανάπτυξη κομμάτια του πληθυσμού να μην μπορέσουν να οδηγήσουν σε έναν αρνητισμό ο οποίος δεν θα είναι τεκμηριωμένος φυσικά. Εμείς λοιπόν έχουμε να κάνουμε πολλά σαν μια Ευρώπη η οποία θα συνεργαστεί και με τους υπόλοιπους σημαντικούς εταίρους σε διεθνές επίπεδο. Με τους ίδιους θόρους θέλω να αναφερθώ στο δεύτερο θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα το μεταναστευτικό. Μιλάμε για ένα θέμα κυρίες και κύριοι όπου η συνεργασία και ο συντονισμός και με τις χώρες προέλευσης και με τις χώρες τράνζιτ και με τις χώρες κατάληξης είναι σημαντικός. Και για την Ισπανία φυσικά αυτό είναι σημαντικό. Από αυτή την άποψη λοιπόν έχουμε ε, ναι, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το έγγραφο που προήλθε ε, από την συνεργασία με το Βασίλειο του Μαρόκου στον τομέα της συνεργασίας και ελέγχου. Εδώ έχουμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο και πρέπει να το θυμίσω. Εμείς απαιτείται να κάνουμε μια νέα προσπάθεια στον τομέα αυτό. Η διάσκεψη του Μαρακές αντιπροσωπεύει, αντιπροσώπευσε τουλάχιστον ένα πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση την πολυμερή της μεταναστευτικής πρόκλησης και η Ισπανία είναι ένας από τους πρώτους που επικύρωσε την πρόταση αυτή. Νομίζω ότι το θέμα αυτό μπορεί να προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα στις κοινωνίες μας σε επίπεδο συζητήσεων. Θα πρέπει ε, να μην γίνεται συζήτηση αποκλειστικά για την παράνομη μετανάστευση, γιατί η τακτική, η νόμιμη μετανάστευση παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε τομείς όπου υπάρχει έλλειψη ανθρώπινων πόρων σε μία Ήπειρο ε, η οποία πολλές φορές χαρακτηρίζεται από την γύρανση του πληθυσμού. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν συνεννοηθούμε με μία άλλη Ήπειρο, την Αφρική, η οποία απαιτείται να περάσει από μία κοινωνικο-οικονομική βαθιά αλλαγή. Αυτός ο πολιτικός δρόμος, ο οποίος έχει μέλλον, ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με όλα τα κράτη-μέλη. Πρέπει να υπάρξει ένας ενιαίος χώρος χωρίς εξωτερικά σύνορα έτσι ώστε να λειτουργήσει σωστά μια κεντρική μεταναστευτική πολιτική. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να μεταρρυθμιστεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χορήγησης Ασύλου και θα πρέπει οι δύο αρχές που θα χαρακτηρίσουν τη δράση μας να είναι η υπευθυνότητα και η αλληλεγγύη. Ε, προφανώς ε, είναι περίπλοκες οι διαδικασίες και οι διαπραγματεύσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα, που κινδυνεύουν. Θα πρέπει να σεβαστούμε και την νομική τάξη της κάθε χώρας. Νομίζω ότι υπάρχουν μερικές φορές βέβαια δράσεις οι οποίες είναι αντίθετες μερικές φορές με τις βασικές ανθρωπιστικές αρχές. Ε, η Ευρώπη δεν πρέπει να ακολουθεί τις μόδες. Η Ευρώπη έχει ένα δημοκρατικό παρελθόν και δημιουργεί τις μόδες. Αυτή είναι και η δύναμή μας και η ισχύ μας. Κύριοι βουλευτέ, ε, η μεγαλύτερη αδυναμία μας εδώ στην Ένωση είναι οι διαιρέσεις μας εποφελούνται, όπως είπα στην αρχή, εκείνοι που θέλουν να αποτύχει το μοντέλο μας. Ένα μοντέλο που βασίζεται σε ένα ε, άρατο κύκλο η δημοκρατία, η πρόοδος και το κράτος ευημερίας. Η υπέρβαση των αδυναμιών μας και των διαιρέσεων μας πρέπει να βασιστεί στην καταπολέμηση των, ε, αυτών των ε, στερεοτύπων. Το Μάη φέτος θα αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη πρόκληση. Ε, έχουμε απέναντί μας ένα μήνυμα που έκανε την Ευρώπη εδώ και δεκαετίες, πριν από λίγες δεκαετίες, ένα πεδίο μαχών. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε με τα δικά μας ιδανικά τις προσπάθειες αυτές. Ε, ποτέ δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένη την ειρήνη, τη δημοκρατία και την ελευθερία. Το είδα με τα μάτια μου όταν ήμουνα στη δεκαετία του 90 στη Βοσνία εργαζόμενο για, τις, ε, για τα Ηνωμένα Έθνη σε μια πόλη που καταστράφηκε από, την, ε, από τον εμφύλιο πόλεμο και το μίσο στο Σαράγεβο. Η, βαρβαρή, η που θεωρούσαμε ότι είχε αποκλειστεί πλέον από την Ήπειρό μα ξαναεμφανίστηκε και τροφοδοτείται από δυνάμεις που πάντα ε, αντιπαραθέτουν το μίσος στην συμβίωση. Δεν απειλούν μόνο την προσπάθεια ενοποίησής μας. Με ε, έμεσο και, και ε, ύπουλο τρόπο αξιοποιούν τα θέματα ορισμένων που λένε ότι είναι αντίθετοι σε αυτές. Παρακαλώ λοιπόν το σώμα σας να μην επηρεάζεται από αυτούς. Απευθύνομαι σε εσά για να είστε αποφασιστικοί στην προστασία των ευρωπαϊκών αξιών και χρειάζεται δύναμη για να αντιμετωπίσετε τις ειρήνες του αυταρχισμού γιατί έχουν ένα μόνο στόχο. Ο στόχος είναι να καταστρέψουν την Ευρώπη. <clears throat> Γι' αυτό κάνω έκκληση σήμερα Υπάρχει αναγκαιότητα να προστατεύσουμε την Ευρώπη, ούτω ώστε η Ευρώπη να προστατεύσει τους πολίτες της. τα επόμενα χρόνια. Είμαι πεπισμένο ότι θα προχωρήσει το κοινό μα εγχείρημα παρά τις δυσχέρειες. Θα έχουμε διαφορές απόψεων, θα έχουμε ε, οπισθοχωρήσεις. Αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι συνολικά θα έχουμε περισσότερη πρόοδο από οπισθοχωρήσεις. Βεβαίως, ε, η πρόοδη αυτή δεν θα βρίσκει τους πάντες σύμφωνους, γιατί αυτό είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε, διότι οι ιδέες μας μπορεί να είναι διαφορετικές, μπορεί και αντιτιθέμενες. Αλλά πρέπει να υπάρχει ε, προσπάθεια να συνδυαστούν αυτές οι ιδέες για να προχωρήσουμε διατηρώντας την ευημερία μας σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει. Ούτως ή άλλως, παρά τις δυσχέρειες, έχουμε μια ε, σταθερή βάση. Την αλληλεγγύη στην πράξη, που αυξάνονται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Το βλέπουμε κάθε φορά που δυστυχώς υπέστημεν τρομοκρατικά χτυπήματα. Είναι, είναι ε, το σπέρμα μιας πραγματικής ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Όταν ένας Ισπανός πολίτης ε, σε αλληλεγγύη με μια τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι βάζει στο σε ένα μέσο κοινωνική δικτύωση μια γαλλική σημαία αγκαλιάζει την ιδέα της Ευρώπης. Και όταν ένας Γερμανός ε, κάνει το ίδιο για την επίθεση στην Βαρκελόνη, αγκαλιάζει την ιδέα της Ευρώπης. Εδώ ξέρουμε ότι υπήρξε μια φρικαλαία επίθεση της, ε, στο Στρασβούργο πριν από ένα μήνα. Όταν εκφράζουμε όλη την αλληλεγγύη μα προ τα θύματα, αγκαλιάζουμε τη σημαία της Ευρώπης. Οι εχθροί της Ευρώπης δεν μπορούν να κάνουν τίποτα ε, έναντι αυτού του αυξανόμενου αισθήματο ε, αόρατη αλλά πραγματική αλληλεγγύη και η οποία εκφράζεται κυρίω μεταξύ των πιο νέων. Αυτοί προβάλλουν την ιδέα τη Ευρώπη ως σύμβολο κατά τη ανισότητα, κατά της αδικίας, κατά του αυταρχισμού, κατά τη φαλοκρατία, κατά του ρατσισμού, για να εκφράσουν απλώ την ε, διαφωνία τους με αποφάσεις που είναι αντίθετες με τη λογική των καιρών και τα συμφέροντά τους. Ε, η... Το να ξεχάσουμε την ιστορία είναι μια ανεπίτρεπτη πολυτέλεια. Δεν μπορούμε να είμαστε διστακτικοί έναντι των ε, ε, αβεβαιοτήτων. Η αποφασιστικότητα θα μας επιτρέψει να επανακτήσουμε το ρυθμό μας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα αυταρχισμό που ζει από μια επινοημένη νοσταλγία. Δεν υπάρχει χειρότερη νοσταλγία από το να νοσταλγούμε κάτι που ποτέ δεν υπήρξε όπως λέει μια, ένα τραγούδι ενός μεγάλου Ισπανού τραγουδιστή. Σε όλες αυτές τις επινοημένες ε, νοσταλγίες ερωτώ, είχαμε σταθερή ειρήνη όταν υπήρχαν ε, κλειστά σύνορα, υπήρχε οικονομική πρόοδος όταν ε, τα τελωνία περιόριζαν τις συναλλαγές, είχαμε περισσότερα κοινωνικά δικαιώματα σε κάθε κράτος όπως τα έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια στα κράτη της Ένωσης πολύ κοντά σε εδώ, στα πεδία μαχών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, θα έχουμε την απάντησή μας. Γι' αυτό σήμερα θέλω να πω ότι έναντι της εσωστρέφειας πρόοδος, έναντι της ρητορική των ε, ε, αποκλειουμένων ταυτοτήτων, θέλουμε ταυτότητες που ε, συμπεριλαμβάνουν τους πάντες. Όπως έλεγε ένα σύντροφος από το Ισπανικό από την Ευρωπαϊκή Σοδημοκρατία ο καταπληκτικό Φρανκ Τίμερμαν, το παρελθόν ποτέ δεν θα είναι το μέλλον για τι κοινωνίε μα. Το παρελθόν είναι ένα. Ε, ένα χώρο που μαθαίνουμε από τι επιτυχίε και τα λάθη μα. Πρέπει να κινητοποιηθούμε για την Ευρώπη. Πρέπει να προστατεύσουμε τι ε, αξίε που κάνουν το εγχείρημά μα ε, ε, μοναδικό στον κόσμο και το οποίο το ζηλεύουν πολύ στον κόσμο. Μόνο έτσι μπορούμε να νικήσουμε αυτού που απ' έξω αλλά και από μέσα προσπαθούν να καταστρέψουν τα ιδεώδη μα. Και θέλουν να το κάνουν, να μην το ξεχνάμε, και θέλω να το υπογραμμίσω και να το θυμίσω. Θέλω να το κάνω για ένα μόνο λόγο. Λόγω των αξιών που υποστηρίζουμε. Που υποστηρίζει η Ένωση. Πρέπει λοιπόν εμεί να απαντήσουμε υποστηρίζοντα αυτέ τι αξίε. Σε αυτή την πορεία, κύριε Βουλευτέ, χρειαζόμαστε πεποίθηση και αποφασιστικότητα. Πρέπει να συνδυάσουμε τα ιδεώδη μα με την προσπάθεια πραγματιστικών λύσεων όπω κάνουμε τα τελευταία 60 χρόνια κοινή ζωή. Το καθήκον μα ω κληρονόμοι αυτή τη μεγάλη κληρονομιά είναι να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε αυτό που κληρονομήσαμε για να το περάσουμε στι επόμενε γενιέ. Εάν μάθαμε κάτι, είναι ότι σε συγκεκριμένε συγκυρίε τη ιστορία μα, όπω αυτήν, το να αντισταθούμε είναι πρόοδο. Σήμερα, στι γενιέ που εσεί εκπροσωπείτε σε αυτό το κοινοβούλιο, ανταποκρίνεται ένα καθήκον: να προστατεύσουμε την Ευρώπη, ούτω ώστε η Ευρώπη να προστατεύσει του πολίτε τη. Ευχαριστώ πολύ. Να προχωρήσουμε τώρα σύμφωνα με το Catch the Eye. Κλείνω το κατάλογο. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη εγγραφεί. Οπότε ζητώ από τους εκπροσώπους των ομάδων να τηρήσουν ε, το χρόνο που τους έχει ήδη κατανεμηθεί. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να ακούσουμε όλους τους συναδέλφους αυτή τη συζήτηση. Παρακαλώ λοιπόν να τηρείτε το χρόνο σας. Πρώτος ομιλητής είναι ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Φραντς Τίμερμανς. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Σάντσες για την πολύ εμπνευσμένη ομιλία του και νομίζω ότι η μία ιδέα που ήθελε να μοιραστεί μαζί μας είναι ότι αν η Ευρώπη θέλει να προστατεύσει τους πολίτες της, εμείς οι πολιτικοί έχουμε συλλογική ευθύνη να προστατεύσουμε την Ευρώπη. Μόνο μια ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες της. Και αυτοί που πολλούν την αυταπάτη ότι μπορεί κανείς να προστατεύσει τους πολίτες απομονώνοντας όσους είναι διαφορετικοί, οικοδομώντας τείχους και φράχτες, πολλώντας ένα ε, απατηλό όνειρο ε, εθνικισμού θα οδηγήσουν στην απογοήτευση, διότι δεν υπάρχει προστασία στον προτεξιονισμό, απομόνωση υπάρχει στον απομονωτισμό και τα έθνη όταν μείνουν μόνα τους στην Ευρώπη δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις πολλές προκλήσεις που μας προσφέρει ο κόσμος. Μόνο μια ενωμένη Ευρώπη μπορεί να κάνει αυτό που απαιτούν οι πολίτες, δηλαδή να τους προστατεύσει και να τους βοηθήσει να διαμορφώσουν το μέλλον τους ως ελεύθεροι και ανεξάρτητοι άνθρωποι. Ξέρω ότι η Ευρώπη ε, υπάρχει στις πλεύρες του ε, Πέντρο Σαντσές, ε, ανήκει στην τελευταία γενιά που μεγάλωσε υπό τη δικτατορία, μια γενιά που μεγάλωσε με το όνειρο της ελευθερίας και η Ευρώπη, η Ισπανία τώρα πια έχει αναλάβει την σωστή της θέση στην καρδιά της Ευρώπης. Το μήνυμα που έχω σήμερα στην κυβέρνηση της Ισπανίας είναι το εξή. Κοιτώντα τα τελευταία 40 χρόνια, νομίζω ότι σωστά μπορούμε να πούμε ότι η Ευρώπη έχει διαμορφώσει την Ευρώπη διότι αυτή ήταν η επιθυμία του ισπανικού λαού. Νομίζω όμως επίσης ότι θα πρέπει να πούμε ότι και η Ισπανία θα πρέπει να συνδιαμορφώσει την Ευρώπη. Χρησιμοποιήστε το δυναμικό σας για να διαμορφώσετε το κοινό μας μέλλον. Είσαστε ισχυροί, ανθεκτικοί και έχετε δείξει στην τρομερή αυτή κρίση που αντιμετώπισε ε, η Ισπανία πώς μπορείτε να ε, την ξεπεράσετε και πιο ισχυρή. Ναι, πράγματι είναι πολύ ε, υψηλή ακόμη η ανεργία. Έχετε σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια όμως. Και νομίζω ότι η αποφασιστικά του ισπανικού λαού αποτελεί έπνευση για όλους μας ε, στην Ευρώπη. Επίσης, ο λαός ε, της Ισπανίας ε, συμμερίζεται τις αξίες ελευθερία, δημοκρατία, ευημερία. Αυτά είναι πολύτιμα πράγματα και δεν θα πρέπει ποτέ να τα θεωρήσουμε δεδομένα. Η Ισπανία έχει σημαντική θέση στην Ένωσή μας και η ευρωπαϊκή της ιστορία πάει πολύ πιο πίσω από το 1985. Ιδιαίτερα όσον αφορά το πόσα χρωστάει η Ευρώπη στην αποφασιστικότητα και τι ιδέε ανθρώπων όπω είναι ο Σαλβαδόρ Ντε Μαδαριάγα που βοήθησε να οικοδομηθεί το ευρωπαϊκό εγχείρημα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ποτέ δεν εγκατέλειψε την ιδέα τη ε, ελεύθερη και δημοκρατική Ισπανία. Και οι άνθρωποι που δεν εγκαταλείπουν τα ιδανικά του ούτε στι πιο σκοτεινέ μέρε είναι αυτοί που μπορούν να διαμορφήσουν με τον καλύτερο τρόπο το μέλλον μα είδε ότι η ταυτότητά μας, ε, η επιτυχία μας ε, είναι συνδεδεμένη του ενός ε, με του άλλου. Τώρα, 40 χρόνια μετά το Σύνταγμα της Ισπανίας, ε, βρίσκεστε στην καρδιά μιας Ενωμένης Ευρώπης η ανάπτυξή σας είναι στο 2%. Η ανεργία ακόμη είναι πολύ υψηλή, αλλά απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν και υπάρχουν πολλά θετικά μηνύματα στην οικονομία. Η οικονομία έχει ορθοποδήσει και πάλι και θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό οφείλεται στο θάρρος και την αποφασιστικότητα των Ισπανών και την αλληλεγγύη της Ευρώπης. Την αλληλεγγύη αυτή την ανταπέδωσε η Ισπανία. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης ε, βοηθήθηκε από την Ευρώπη, αλλά έχει δείξει επανειλημμένα ότι ε, δείχνει καθημερινά την αλληλεγγύη τη με το υπόλοιπο τη Ευρώπη. Το βλέπουμε αυτό στο θέμα τη μετανάστευση. Η Ισπανία και η Μάλτα, ακόμη και σε πολύ δύσκολου καιρού, ε, επιδεικνύουν αλληλεγγύη απέναντι σε ανθρώπου που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. εσύ ήσουν ηγέτης, καλωσόρισες εσύ τους, ε, ε, ε, τους ναυαγούς στο πλοίο Aquarius. Στο όνομα το, του ισπανικού λαού είπες ότι δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να πνιγούν. Αυτό είναι πραγματική πολιτική ηγεσία. Δεν επέλεξες τον εύκολο δρόμο, δεν έστρεψες αλλού το βλέμμα, δεν κατηγόρησες του ε, ε, πρόσφυγες απλά ανέλαβε την ευθύνη για τη μοίρα τους. Ε, οι εικόνες των πλοίων αυτών και οι διαιρέσεις που ε, δημιούργησαν ακόμη και οι λίγες αφήξεις στις ακτές μας έδειξαν τις δυσκολίες και τώρα θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το κοινό σύστημα ασύλου. Μόνο με μεταρρυθμίσεις θα μπορέσουμε να έχουμε μια βιώσιμη λύση. Μόνο η προστασία των συνόρων δεν αρκεί. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ασύλου που να βασίζεται στην αλληλεγγύη και στι θεμελιώδει αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα επίση, Πέδρο, να τονίσω αυτό που είπε για την Αφρική. Εάν υπάρχει μία ήπειρος που θα καθορίσει το μέλλον της Ευρώπης. Αυτή η Ήπειρος είναι η Αφρική. Κανείς άλλος στον κόσμο δεν μπορεί ή δεν θέλει να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Είναι η ε, αδερφή Ήπειρός μας. Ε, απέχει πολύ λίγο από τις ακτές μας και εάν δεν αναλάβουμε κοινή ευθύνη, συλλογική ευθύνη για το μέλλον και των δύο υπήρων, τότε τα προβλήματα της Αφρικής ε, δεν θα μπορέσουμε να τα κρατήσουμε μακριά από την Ευρώπη όσο υψηλούς φράχτες και να χτίσουμε. Χρειάζεται ένα μέλλον στο οποίο να μπορούν να πιστέψουν οι άνθρωποι της Αφρικής. Χρειαζόμαστε σταθερότητα στην Αφρική, ώστε και η Ευρώπη να είναι σταθερή και ελεύθερη στο μέλλον. Πέδρο, σε καλό να οδηγήσει την Ευρώπη ώστε να καταλάβει ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο των μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου και αν βρίσκονται. Στον προϋπολογισμό μας θα έχουμε σχεδόν ε, τριπλάσια αύξηση, 33 ε, ε, δισεκατομμύρια ευρώ για τα θέματα μετανάστευσης. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη, όχι μόνο επειδή για την Ισπανία, όχι μόνο επειδή έχετε επιδείξει το, τόση αλληλεγγύη, αλλά επειδή γνωρίζετε και τις, επειδή έχετε δει τρομερές τρομοκρατικές επιθέσεις στο έδαφος της. Με 9 δισεκατομμύρια ευρώ θα στηρίξουμε και τον ε, ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης σε κάτι το οποίο θα, προωθήσει, θα βοηθήσει την ανάπτυξη της ισπανικής οικονομίας. Ε, επίσης, ε, πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν ε, κινητοποιηθεί με το ε, σχέδιο Juncker και έτσι έχουν βοηθηθεί ε, περίπου 45.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και είδαμε δημιουργία θέσεων εργασίας και στήριξη της κυκλικής οικονομίας στην Ισπανία. Κύριε Πρωθυπουργέ, γνωρίζω την προσήλωση της χώρας σας στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και ε, πρέπει και η Ισπανία και η Ευρώπη να εφαρμόσει αυτόν τον μετασχηματισμό και θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία να χαιρετήσω τον συνάδελφό μου που κάθεται εδώ δίπλα μου που έχει φροντίσει σε όλο τον κόσμο ε, έχει καταβάλει προσπάθειες ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να πετύχει τους στόχους του Παρισιού. Νομίζω ότι έχει ηγηθεί παγκοσμίω στο θέμα αυτό και ε, του αξίζει η αναγνώρισή μας και η εκτίμησή μας. Το νέο πρόγραμμα InvestEU ε, έχει τη δυνατότητα ε, να κινητοποιήσει επιπλέον 650 δισεκατομμύρια ε, ευρώ για επενδύσεις ανάμεσα στο 2021 και το 2027. Επίσης θα υπερδιπλασιαστεί η χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Erasmus και είχα τη χαρά να ε, εργαστώ και στο παρελθόν ε, με τον δημιουργό του ε, προγράμματος Εράσμους. Πραγματικά πρόκειται για πολύ ισχυρό πνεύμα. Ο Χουάν Μαρίν είναι ο άνθρωπος αυτός. Και έχω δει πολλούς ε, νέους ανθρώπους ε, των οποίων ε, οι γνώσεις και το ανοιχτό πνεύμα έχουν εντυπωσιάσει όλους μας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μπορέσουμε σύμφωνα να συμφωνήσουμε πάνω στο νέο προϋπολογισμό και βασίζομαι στην υποστήριξη του Πέντρο, των ομολόγων του και του Κοινοβουλίου για να το πετύχουμε αυτό. Θα ήθελα να τονίσω την αξία, την ποιότητα του θεματολογίου της Ισπανικής κυβέρνησης. Χρειαζόμαστε ένα καλύτερο σχέδιο για να κλείσουμε την ψαλίδα αμοιβών ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη. Ε, θα πρέπει να κλείσουμε την ψαλίδα στις ε, συντάξεις ε, που ανέρχεται σε 40% στην Ευρώπη. Θα πρέπει να σπάσουμε τη γυάλινη οροφή, να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες της Ευρώπης. είναι απαράδεκτη η κατάσταση αυτή τη στιγμή και βασίζομαι στην κυβέρνηση του Πέντρο για για να ε, το πετύχουμε αυτό. Γιατί δεν έχουμε δώσει τέλος στη βία ει βάρος των γυναικών. Είναι υποχρέωσή μας αυτό, είναι καθήκον μας. Και γιατί δεν ονοματίζουμε αυτούς που ε, εσφαλμένα επικαλούνται οικογενειακές αξίες ε, για να στερήσουν από τις γυναίκες τα πλήρη δικαιώματα. Ε, δεν επιτρέπεται να δικαιολογούμε τη βία ε, στο, ε, σε ένα γάμο, στο οικογενειακό πλαίσιο. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, κύριε Πρωθυπουργέ, η Ισπανία και η ευρωπαϊκή της ιστορία αποτελούν υπόδειγμα για την Ευρώπη. Δείχνει τι σημαίνουν οι αξίες για τις οποίες μιλάμε και δείχνει τι μπορούμε να πετύχουμε με τη συνεργασία και με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Η Ευρώπη προστατεύει, αλλά πρέπει και εμεί να προστατεύσουμε την Ευρώπη. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Ο πρώτος ομιλητής εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων είναι ο επικεφαλής του ΕΛΚ, ο κύριος Μάνφρετ Βέμπερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, καλώς ήρθατε η παρουσία σας εδώ δίνει μια μεγάλη όθηση για το 2019, γιατί εσείς είστε φιλοευρωπαϊστής, ε, ξεκάθαρα δεσμευμένος σε ευρωπαϊκούς ε, στόχους. Γι' αυτό είναι θαυμάσιο που σας έχουμε εδώ. Η Ευρώπη σημαίνει για την Ισπανία ειρήνη και ευημερία. Η Ισπανία σημαίνει για την Ευρώπη ισχύ, φρέσκες ιδέες και ηγεσία. Γι' αυτό είναι πολύ καλό που σας έχουμε εδώ. Από την άλλη, είναι σημαντικό γιατί το 2019 είναι το έτος όπου θα εορτάσουμε τη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ευρωπα... ευρωεκλογέ θα λάβουν χώρα. Και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για τη δέσμευσή σα όσον αφορά την υποστήριξη του Φραντς ε, Τίμερμαν ως σοσιαλιστή υποψηφίου είναι μια σαφής ένδειξη ότι πιστεύετε στη δημοκρατική ιδέα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα το κρατήσετε ζωντανό, ε, θα κρατήσετε ζωντανή αυτή την αρχή και μετά τις ευρωεκλογέ. Όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης, ε, δυστυχώς θα πρέπει να μιλήσουμε και για εθνικισμό και ρατσισμό. Έχουμε τα χθεσινά αποτελέσματα των εκλογών. Ε, ε, ε, οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι βρίσκονται στο ίδιο πλοίο σύμφωνα με το πνεύμα των ιδρυτικών πατέρων της Ευρώπης. Οι ευρωπαϊκές αξίες βρίσκονται σε κίνδυνο. Οι εξτρεμιστές δεν έχουν χρώμα. Εσείς είστε ένας φιλοευρωπαϊστής, αλλά η κυβέρνησή σας δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς την υποστήριξη των ε, ακραίων ε, αριστερών και των ε, εκείνων που είναι υπέρ της απόσχησης. Ο στόχος όμως της Ευρώπης είναι να υπάρξει σταθερότητα και, να... και ο Φραντς Τίμερμαν εξήρε την θετική εξέλιξη της ισπανικής οικονομίας ε, τα τελευταία έτη μετά την οικονομική κρίση. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω σε όλους, αυτό έγινε χάρη στις προσπάθειες της κυβέρνησης του Μαριάνο Ραχώη να δημιουργήσει προποθέσεις για αυτή την ε, οικονομική επιτυχία της Ισπανίας. Και τώρα εσείς ε, θέλετε να πάρετε πίσω τις μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας που έκανε ο Μαριάνο Ραχώη. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό θα ήταν το εσφασμένο μήνυμα όσον αφορά τη δημιουργία ενός οικονομικού μέλλοντος για την Ισπανία αυτό προποθέτει να κάνει κανεί μεταρρυθμίσει. Ε, μεταρρυθμίσεις, Η Ευρώπη θέλει να αυξήσει τα έσοδα των εργαζομένων. Άρα λοιπόν παρακαλώ να διατηρήσετε τι μεταρρυθμίσει, μην ακούσετε του λαϊκιστέ. Δεύτερον, ε, σεβόμαστε πάρα πολύ την κυβέρνησή σας, έστω και αν δεν συμμεριζόμαστε τις ίδιες ε, πολιτικές αξίες και ιδέες αλλά μας ανησυχεί το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας. Αυτή τη στιγμή δεν ε, πετύχατε μια επικοδομητική πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο για το προϋπολογισμό που παρουσιάσετε. Ωστόσο, εκπροσωπείτε μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες στην Ευρωζώνη και μια τέτοια μεγάλη οικονομία χωρίς ε, προεπολογισμό ε, οδηγεί σε αστάθεια. Και αυτό ε, και με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αστάθεια στην Ευρώπη. Τώρα, όσον αφορά τη μετανάστευση, εμεί στο και έχουμε ξεκάθαρε προτεραιότητε. Ε, το σχέδιο Μάρσαλ για την Αφρική, ένα φιλόδοξο πλάνο επαναγκατάσταση των προσφύγων. Θέλουμε να βοηθήσουμε του πρόσφυγε από τη Συρία και άλλε περιοχέ. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι η παράνομη μετανάστευση θα πρέπει να τερματιστεί. Θα πρέπει ε, να καταστρέψουμε το, να πατάξουμε το απάνθρωπο μοντέλο παράνομης ε, μετανάστευσης των διακινητών. Και εδώ η Ισπανία ε, φέρει ένα μερίδιο ευθύνη. Ε, τα παράνομα περάσματα από την Ισπανία έχουν διπλασιαστεί ε, τον τελευταίο χρόνο. Ακούω πολύ συχνά το επιχείρημα ότι είναι δύσκολο να προστατευτούν τα σύνορα. Εγώ ε, πέρσι το καλοκαίρι πήγα στην άλλη πλευρά της Υπήρου, στα σύνορα μεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας. Και εκεί φτιάχτηκε ένας φράχτης ύψους ενός ε, μέτρου για 100 χιλιόμετρα. Και αυτό μας δείχνει ότι αν υπάρχει πολιτική βιβούλεση μπορεί να προστατευτούν τα σύνορα ε, και τέτοια μέτρα ε, όπως ε, τέτοιος φράχτης είναι αποτελεσματικά. Εάν θέλουμε να πατάξουμε τον εξτρεμισμό θα πρέπει να προστρέξουμε σε τέτοια μέτρα και αναμένουμε από την Ισπανία να προστατεύσει τα σύνορα όπως στην Χάουτα και στη Μελίγια. Στην Ισπανία ε, υπάρχει και ένα πρόβλημα με τις απασχεστικές στάσεις στην ε, Καταλωνία. Εμείς ως ΕΛΚ στηρίζουμε την και αικαιρότητα της Ισπανίας και στηρίζουμε την κυβέρνηση όσον αφορά την διατήρηση της ενότητας της Ισπανίας. Η Ευρώπη έχει κονδομηθεί επί της αρχής του κράτους ε, δικαίου, τα ίδια και η Ισπανία. Και αυτό έπραξε και η κυβέρνηση Ραχώ και εμείς θα σας υποστηρίξουμε εάν θέλετε να προσφέρει στις ίδιες αρχές. Η δική μου πολιτική ομάδα ε, υπερψήφισε ένα κομμουνιστή αντιπρόεδρο, αλλά δεν θέλαμε να υπερψηφίσουμε έναν ακροδεξιό υποψήφιο, γιατί θέλουμε να εγγυηθούμε οι εθνικιστές να μην έχουν λόγο για το μέλλον της Ευρώπης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Έχετε πολλά πράγματα να κάνετε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της πολιτικής μας ομάδας και να σας ευχαριστήσω και για την ε, ε, βούλησή σας Ισπανίας ε, ε, όσον αφορά τις φιλοευρωπαϊκές ε, αρχές στην Ευρώπη. Όχι εθνικισμοί, αλλά ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Σας ευχαριστούμε για την συνεισφορά σας. Τώρα ουρουλάτη in aula. Serve sempre il veterinario. Prossimo intervento è quello Επόμενη ε, παρέμβαση του κυρίου Ούντο Μπούλμαν. Αγαπητέ Πρόεδρε της Κυβέρνησης, αγαπητέ Πέδρο, καλώς όρισες ε, στο Ευρωκοινοβούλιο. Αγαπητέ Πέδρο. I, cannot help. I cannot Αγαπητέ Πέδρο, δεν μπορώ παρά να αναφέρω τα λόγια σου. Αν η Ευρώπη πρέπει να μας προστατεύει, Πρέπει εμείς να προστατεύσουμε την Ευρώπη. Μακάρι να ήταν αυτό το σύνθημα όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Μακάρι να ήταν αυτό το σύνθημα όλων των Ευρωπαίων ηγετών και να αποτελεί το ορόσημο ε, έναντι το οποίο θα πρέπει να μετρηθεί οποιοδήποτε ε, με πολιτικές ευθύνες στην Ευρώπη. Δυστυχώς είμαστε πολύ μακριά από αυτό και γι' αυτό και σε περιμέναμε με ανυπομονησία. Θέλαμε να σε ακούσουμε αυτή την εμπνευσμένη και παθιασμένη ιδέα της ε, δικαιοσύνης και της πρόοδου για την Ευρώπη μας. Δυστυχώ δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά, συνάδελφε κύριε Βέμπερ, όπω το παρουσιάζετε. Όλοι βρισκόμαστε στο ίδιο σκάφο, αλλά εάν θέλουμε να πατάξουμε τον εθνικισμό, αν θέλουμε να παρεμποδίσουμε ότι η Ευρώπη να μην γίνει το θύμα των ακροδεξιών, τότε θα πρέπει το σκάφος αυτό να έχει και μια κατεύθυνση πλεύσης, θα πρέπει να αναπτύξει ένα δυναμισμό και θα πρέπει να εμποδίσουμε την τελμάτωση των, τις δεκαετία όπου οι άνθρωποι στην Ευρώπη περιμένουν να παράσχουμε αποτελέσματα και να τις προστατεύσουμε όσον αφορά την κοινωνική τους κατάσταση, τις συντάξεις, τις προεπτικές στο σύγχρονο κόσμο εργασία. Και αυτό είναι το ουσιαστικό πρόβλημα. Ότι όλοι λένε ότι βρίσκονται στο ίδιο σκάφο, αλλά κανεί δεν μπορεί να αναπτύξει τον δυναμισμό μέσω του οποίου μπορεί κανεί να νικήσει τα κύματα και να πλεύσει εν μέσω των απειλών και των κινδύνων σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί από την άλλη πλευρά κάθεται κάποιο σαν τον Πούτιν, ο οποίο δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τι δικέ μα ιδέε ελευθερία. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι από την άλλη υπάρχει και ο Τραμπ, ο οποίο δεν έχει ιδέα για την ε, δυνατότητά μας να οργανώσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη στην κοινωνία μας. Και τι περιμένουμε λοιπόν, γιατί δεν ε, μπορούμε να πυροδοτήσουμε αυτό το δυναμισμό ε, στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Εμένα μου άρεσαν τα όσα είπε ο Πέδρο Σάντσεθ, γιατί εκπροσωπούν ένα πρόγραμμα ε, κοινή ε, καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης στο υπόβαθρο των ανησυχιών που έχουν οι πολίτες της Ευρώπης. Θα πρέπει να αντλήσουμε το δίδαγμα, να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, να έχουμε αποτελέσματα. Ο Πέτρος Σάντσεθ ε, το εξέφρασε αυτό στην ομιλία του. Αυτό χρειαζόμαστε τα επόμενα χρόνια της νέας εντολής. Και θα, θέλω να είμαι ειλικρινής. Μου άρεσε γιατί ε, αυτά υπόθηκαν από τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας μιας ε, χώρας και θέλω να τονίσω αυτό το οποίο είπε ο Φραντ όπου η μοίρα της Ευρώπης ε, έχει, ε, συγκαθορίζεται. Μία χώρα με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, ε, η οποία, μια χώρα η οποία γνωρίζει τις διαφορετικές ρίζες της. Μια χώρα όπου μπόρεσε να νικήσει το φασιστοειδές καθεστώς του Φράγκο μια χώρα που δεν θέλει να ξαναβυθιστεί στην εποχή της κατάργησης της δημοκρατίας και του ζώφου. Ε, στην Ισπανία και ξέρουμε ότι είναι σε καλά χέρια. Το πρόγραμμα το οποίο μας παρουσίασε ο Πρωθυπουργό είναι πρόγραμμα το οποίο η δική μου πολιτική ομάδα θεωρεί ότι απηχεί τις αξίες της. Είπαμε ότι δεν θέλουμε να μιλάμε πλέον για την οικονομία χωρίς την προεπτική της απασχόλησης των κατοίκων, των ε, πολιτών, αλλά δεν μπορούμε ε, να μην αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μία αλλαγή παράλληλα η οποία θα σώσει τον πλανήτη. Αλλά αυτή η αλλαγή θα πετύχει μόνο εφόσον πάρουμε τους πολίτες με το μέρος μας. Μόνο εφόσον τους δώσουμε ελπίδες και προοπτικές. Δεν μπορεί να είναι μία αλλαγή η οποία να είναι εναντίον των πολιτικών. Δείτε την εμπειρία της Γαλλίας, την εμπειρία του Μακρόν. Πρέπει να ενισχύσουμε τους πολίτες ούτω ώστε να σταθούν στο πλευρό μας αυτή την αλλαγή. Γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική προοπτική, να της δώσουμε ένα αναθέσουμε στα επίκεντρα της πολιτικής μας. Ε, ναι, Βεβαίω ε, το διακύβημα είναι το πώς ε, γίνεται η διακυβέρνηση ε, και το μήνυμα από τη Μαδρίτη, το γεγονός ότι πετύχατε, Πέδρο Σάντσεθ, να φτιάξετε μια έξυπνη κυβέρνηση όπου πραγματικά μπορούν ε, υπουργοί με υψηλές δεξιότητες να συνενώσουν τις δυνάμεις της. Έχετε μια επίτροπο βιωσιμότητας και επιτέλους ένα ξεκάθαρο μήνυμα όχι μόνο για την ισότητα των δύο φύλων αλλά ε, να ε, προωθήσετε γυναίκες με υψηλά προσόντα στην κυβέρνησή σας. Θα ήθελα να σας συγχαρώ. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, μιλήσατε για το μέλλον της Ευρώπης και πολύ σωστά την ομιλία σας την συμπληρώσατε με τις ιδέες σας για το Brexit. Ο Αντιπρόεδρος Τίμερμαν σε ευχαρίστησε τους ε, Βρετανούς στρατιώτες που απελευθέρωσαν τη χώρα του από τους Ναζί. Εγώ είμαι Γερμανός, ο πατέρας μου. Ε, πέθανε στον πόλεμο, σκοτώθηκε στον πόλεμο και το ε, σπίτι μας βομβαρδίστηκε το 1943 και χάσαμε την μάχη της Βρετανίας. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό, αλλά θα ε, λυπηθώ πάρα πολύ εάν χάσουμε τη μάχη που δίνουμε τώρα υπέρ της Βρετανίας. Το Brexit είναι μια κατάσταση από την οποία θα χάσουν ε, και η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι οικονομικά, πολιτικά και ηθικά ε, θα χάσουν. Οικονομικά διότι το Brexit θα αντιστοιχούσε ε, στο να αποχωρήσουν 19 χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενιαία αγορά ταυτόχρονα. Πολιτικά, διότι, η, ε, διότι το Ηνωμένο Βασίλειο πάντα ήταν η φωνή της λογικής, ε, της επικουρικότητας, της αποκέντρωσης κλπ. Και ηθικά, διότι όπως είπαν προηγουμένως και πολύ σωστά διάφοροι ευρωβουλευτές, από το Brexit θα γίνουμε όλοι φτωχότεροι. Οι προηγούμενες συζητήσεις δείξαν ότι σχεδόν όλοι ε, λυπούνται για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, εκτός από τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ στα αριστερά μου, αλλά ούτε ένας δεν έχει προσφέρει μια λύση για να σταματήσει το Brexit και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γίνει αυτό. Ε, πάνω από 140 μέλη του Ευρωκοινοβουλίου απευθύνθηκαν ε, στον ε, λαό της Βρετανίας, ε, τους ζητάνε δεύτερο δημοψήφισμα. Συμφωνώ με αυτό, αλλά θα έπρεπε αυτό να έχει γίνει νωρίτερα, διότι σε αντίθεση με αυτό που είπε ο κύριος Φερχόφστατ, δεν είναι το πρόβλημα μόνο οι διαμάχες εντός του συντηρητικού κόμματος. Υπήρχαν λόγοι που το Ηνωμένο Βασιλιά να σκέφτεται την Ευρώπη. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας μιλούσαμε για την επικουρικότητα, αλλά τι έγινε, ε, συγκέντρωση τη εξουσία. Μιλούσαμε για ανταγωνισμό, βλέπουμε όμω όλο και περισσότερη εναρμόνιση. Μιλούσαμε στη συνθήκη της Λισαβόνας ε, για την ε, ευθύνη κάθε κράτους για το χρέος του, αλλά τελικά τι κάνουμε, κοινωνικοποιούμε το χρέο. Ήρθε η ώρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αρχίσουν να κάνουν άλλα πράγματα. αναφέρθηκε μια νέα συμφωνία ώστε η ΜΕΗ να συγκεντρώσει την πλειοψηφία εντός του Κοινοβουλίου της. Αλλά ας ε, κάνουμε ε, κάτι άλλο. Ας δώσουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο μια ε, συμφωνία που θα, την, το κάνει να θέλει να παραμείνει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνούμε ότι έχουμε ευθύνη για το Brexit. Ας προσφέρουμε λοιπόν μια νέα συμφωνία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να παραμείνει εντός του της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό μπορεί μόνο να είναι μια ειδική ε, προσωρινή συμφωνία για τη μετανάστευση. Αντί πάντα να κατηγορούμε τη Βρετανία, ας αναγνωρίσουμε ότι η Ευρώπη και οι Βρυξέλλες αποτελούν μέρος του προβλήματος. Θα πρέπει να γίνουμε όμως μέρος της λύσης. Ας ε, αγωνιστούμε για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ. Εξ το φίλο, ελευθέρων, ο κύριο Φερχόφστατ. Μάλιστα, τέσσερα λεπτά, γιατί έχω έναν Ισπανό, έναν Καταλανό και έναν Βάσκο συνάδελφο που θέλουν να πάρουν το λόγο μετά από μένα και τη θέλω τη ζωούλα μου ακόμη. Ε, Ένα χαρακτηριστικό της Ισπανίας ε, και εσείς είστε ζωντανή απόδειξη αυτού είναι πως ίσως είναι Είστε η πιο ε, φιλοευρωπαϊκή χώρα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, γιατί έχει το θάρρος να μιλά για Ομοσπονδιακή Ευρώπη. Πολλοί από τους συνάδελφούς σας που ήρθαν εδώ δεν είχαν αυτό το θάρρος. Δεν είναι τυχαίο, πιστεύω αυτό. Πιστεύω διότι η ευρωπαϊκή ιστορία και η ισπανική δημοκρατία είναι αλληλένδετες. Πιστεύω επίσης επειδή τα, τελευταίες δεκαετίες ε, το Υπουργείο Εξωτερικών σας και μέλη εδώ σε αυτήν την, ε, την, την ε, ολομέλεια ο Μέντες Δεβίγκο, η Παλάσιο, ο Μιγγέλ Μορατίνος που ήταν πρώην ε, υπάλληλο και τέλος υπάρχει ανταγωνισμός στην ισπανική πολιτική ώστε να, ποιος θα είναι ο πιο φιλοευρωπαϊστής από τα κόμματα σας ανάμεσα στο ΠΕΠΕ, το ΨΟΕ και τους Σιουταδάνους και πολύ μου αρέσει αυτό να βλέπω και θα ήθελα σε κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει αυτού του είδους η άμυλα. Ποιος θα είναι ο πιο φιλοευρωπαϊστής δηλαδή ανάμεσα στα κόμματα. Αλλά πρέπει να σας πω, δεν ξέρω, είναι η 15η συζήτηση που κάνουμε για το μέλλον της ε, Ένωσης και λίγο αισθάνομαι μια... Έχω μπερδευτεί γιατί κάθε φορά έρχεται ένας πρόεδρος, έρχεται ένας Πρωθυπουργό, κάνει ένα ολόκληρο κατάλογο των νέων ευρωπαϊκών πολιτικών που πρέπει να κάνουμε, κοινωνική πολιτική, φορολογική πολιτική, μεταναστευτική πολιτική, ευρωπαϊκό στρατός και ποτέ δεν λέμε γιατί δεν το κάνουμε στην πράξη. Ποιο είναι το εμπόδιο, γιατί πάντοτε ενεργούμε πολύ λίγο και πολύ αργά σε σύγκριση με τους Αμερικανούς, ας πούμε, που σε 9 ε, μήνες ε, ε, τα κατάφεραμε την κρίση και εμείς μετά από 9 χρόνια δεν έχουμε ακόμα τραπεζική ένωση. Τεράστια τραγωδία στη Μεσόγειο και σας συγχαίρω ε, ε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσατε τους πρόσφυγες του Ακουάριου. Αλλά ας είμαστε ειλικρινεί, αυτή είναι η συνέπεια ε, της απάνθρωπης ε, νασιοναλιστικής, εθνικιστικής δηλαδή πολιτικής του Σαλβίνη. Ε, και είναι και λόγω της έλλειψης ευρωπαϊκής πολιτικής. Γιατί δεν έχουμε ακόμα τέτοια ευρωπαϊκή πολιτική, γιατί ακόμα δεν έχουμε συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου, για παράδειγμα, μετά από τόσο πολλά χρόνια τραγωδιών στην Μεσόγειο. Γιατί δεν έχουμε ευρωπαϊκό στρατό ήδη σήμερα, γιατί ακόμα αγωνιζόμαστε με τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης, εννέα χρόνια μετά από την αρχή της κρίσης. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα για μένα και ελπίζω ότι στην απάντησή σας σε λίγα λεπτά θα μας μιλήσετε για αυτό το πρόβλημα. Για μένα το πρόβλημα είναι ότι έχουμε κακούς θεσμούς αυτή τη στιγμή στην Ένωση και οι καλοί θεσμοί οδηγούν σε κακά αποτελέσματα. Ενώ οι καλοί θεσμοί καλά αποτελέσματα. Το πρόβλημα είναι και θέλω να το επαναλάβω και θα το επαναλαμβάνω συνέχεια μαζί με κάποιου από εσά. Είναι ο κανόνας της Ομοφωνία που ισχύει στην Ένωση και ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είναι το βασικό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αποφασίζει με την πλειοψηφία και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που εξακολουθεί να αποφασίζει με την ομοφωνία. Όλα τα παραδείγματα που σας έδωσα, όλα αυτά τα πέντε ζητήματα είναι μπλοκαρισμένα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σας κάνω λοιπόν έκκληση τώρα και στα επόμενα χρόνια να δώσετε αυτή την πολιτική μάχη που πρέπει να δώσουμε γιατί διαφορετικά θα μείνουμε σε ευχολόγια που ποτέ δεν θα υλοποιηθούν. Και κύριε Πρόεδρε, πρώτη φορά έκανα κάτι αδύνατον μόλις έμεινα στα τέσσερα λεπτά μου κύριε Πρόεδρε. Ναι, η κυρία Κέλλερ για τους ε, πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ για την ομιλία σας. Πιστεύω ήταν πολύ φιλοευρωπαϊκή και ισχυρή και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί πολλοί ανησυχούν όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης, πολλές ε, κυβερνήσεις ε, αποτυγχάνουν στην εξασφάλιση του κράτους δικαίου και της δημοκρατία στη χώρα τη. Άρα είναι θετικό το ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε τα πράγματα μπορεί να γίνουν διαφορετικά. Αυτό είναι πολύ καλό. Και θα ήθελα να συγχαρώ επίση για όλα τα μέτρα τα οποία λήφθησαν στην Ισπανία και που αντανακλούν ακριβώ τι δεσμεύσει που εξφράσατε εδώ και την απόφαση σα, για παράδειγμα, να αυξήσετε τον ελάχιστο μισθό ε, των 900 ε, ευρώ. Κάτι που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολλέ οικογένειε. Επίση, συνδυασμό με με, με, τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος που είναι μια μεγάλη βελτίωση. Εμείς επιθυμούμε μια κοινωνική Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες στο Συμβούλιο και στις χώρες μέλη και ελπίζω και άλλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά σα. Και δεύτερον, η απόφασή να εξασφαλίσετε ε, η, τα νοικοκυριά να βάλουν ε, ε ηλιακό, ηλιακές ε, στις στέγες τους. Ε, ε ούτως ώστε ο καθένας ε, μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια διάσωσης του πλανήτη. Χρειαζόμαστε αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα. Επίσης, ε, χάρηκα, γιατί όπως επαναφέρατε, η κυβέρνησή σας έχει το υψηλότερο ποσοστό γυναικών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα και απέχουμε πάρα πολύ από μια ε, δρέωση της όντας των φίλων. Θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες γιατί Υπάρχουν ε, πολλέ χώρε που παραβιάζουν τα δικαιώματα των γυναικών και είναι πολύ θετικό να υπάρχουν κυβερνήσει που προωθούν μια φιλόδοξη ε, ατζέντα που είναι υπέρ τη ισότητα των φύλων. Βεβαίω, το έργο είναι δυσχερέ, κληρονομήστε πάρα πολλά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι η κατάσταση στην Καταλωνία. Ε, και, και ο προκάτοχός σας υπήρξε εξαιρετικά αδιάλακτος. Τώρα έχετε εσείς το θέμα στο τραπέζι σας και είναι ξεκάθαρο ότι μόνο μια δημοκρατική πολιτική λύση θα μπορούσε να οδηγήσει την Ισπανία μπροστά και περιλαμβάνει επίσης μια λύση και για τους φυλακισμένους, επίσης τα πρώην μέλη της δικής μας πολιτικής ομάδας που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις φυλακές. Ε, Χρειάζεται λοιπόν να ξεκινήσει ένας ειλικρινής διάλογος, γιατί μόνο με μια θετική βούληση και από τις δύο πλευρές ε, θα έχουμε αποτελέσματα και θα έρθουμε πιο κοντά σε μια λύση που χρειάζεται κατεπηγόντως για την Καταλωνία, για το σύνολο της Ισπανίας και για ολόκληρη την Ευρώπη. Αναφέρεται και η Πρωθυπουργέ τις Ευρωπαϊκές Αξίες και εδώ υπάρχουν κάποιες ανησυχίες όταν βλέπουμε την κατάσταση στην Ανδαλουσία και το σχηματισμό της τοπικής κυβέρνησης εκεί. Γιατί ένα ακροδεξιό εξερμιστικό κόμμα θα συμπεριληφθεί στην κυβέρνηση. Γίνεται ανεκτό και λυπούμε που η συντηρητική και οι δεξί συμφωνούν γι' αυτό. Και ε, είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς συμμερίζονται αυτές τις ανησυχίες και δεν ε, χαίρονται για αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναλυφθεί συγκεκριμένη δράση. Όλες οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να προσπαθήσουν να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί πραγματικά είναι επονίδη συμφωνία όταν μια πολιτική ομάδα δέχεται να συνεργαστεί με ένα ακροδεξιό κόμμα. Εμείς ε, υποστηρίζουμε τις γυναίκες που αυτή τη στιγμή δηλώνουν για την ισότητα των φίλων γιατί η βία κατά των γυναικών δεν έχει καμία θέση οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι πολλοί από τους στόχους που αναφέρατε, ισότητα των φύλων, κοινωνική Ευρώπη κλπ. Όλα αυτά προποθέτουν το ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα λοιπόν ελπίζουμε ε, τις δικές σας πρωτοβουλίες στο Συμβούλιο, να ε, στηρίξετε το Συμβούλιο σε αυτή την κατεύθυνση και να εξασφαλίσετε οι συνάδελφοι στο Συμβούλιο επίσης να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση μιας σοσιαλιστικής και φιλοδημοκρατικής ε, Ευρώπης. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της κυρία Βερμέχου. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Τσάντσες, θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ παρόν και για το ότι συμβάλλεται στην ευρωπαϊκή συζήτηση που είναι ε, πιο απαραίτητη από ποτέ ενώπιον ε, της ε, ανάδυσης των, ακροδεξιών δυνάμεων και στην Ισπανία. Ωστόσο, δεν μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα με τους για την διάγνωσή σας με τις λύσεις που δίνεται σε όλους αυτούς τους κινδύνους που έχουν αναδεθεί. Σε σχέση με την ακροδεξιά, αυτά τα σχήματα φασιστικών τάσεων θα πρέπει να τι αντιμετωπίσουμε και να τις ε, κόψουμε από τη ρίζα. Αυτά τα φαινόμενα στην ουσία ε, οφείλονται στις ε, περικοπές που έχουν κάνει πολλές κυβερνήσεις ε, έναντι των εργατικών τάξεων. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές έχουν μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το κράτος πρόνοιας και η διαχείριση της κρίσης είναι και αυτή υπεύθυνη για μια αβάσταχτη ανισότητα. Με τις πολιτικές στην υπηρεσία των προνομιούχων ε, έχετε προκαλέσει μια, ένα μεγάλο κοινωνικό ε, πόνο και μια κοινωνική κρίση και η Ισπανία συμμετείχε στις πικρές αυτές ε, στιγμές που ζούμε. Η συνταγματική μεταρρύθμιση εξπρέση και οι περικοπές στην παιδεία, στην υγεία, στις συντάξεις, ε, δύο εργατικές ε, μεταρρυθμίσεις ιδιαίτερα ζημιογόνες για τους εργαζόμενους. Είναι κάτι που δεν μπορεί να ξανασυμβεί. Αυτά όλα δημιούργησαν το, κατάλληλο λίπασμα, το κατάλληλο έδαφος ώστε η ακροδεξιά να εκμεταλλευτεί την απελπισία της κοινωνίας κοινωνικής και να παρουσιάσει ψευδείς ε, εχθρούς και ψευδείς λύσεις. Ε, κύριε Σάντσε, η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα έχει πάνω από 140 εκατομμύρια φτωχού και επισφαλεί εργαζόμενου. Συνέπεια και αυτό τη ε, εδαφική ασυμμετρία του παραγωγικού μοντέλου, μέσω του οποίου ζημιώνεται το, ο νότο τη Ευρώπη. Μα καταδικάζουν σε υποβοηθούμενα μοντέλα που βασίζονται σε, χα, σε χαμηλά αμοιβόμενα εργατικά χέρια θέσεις επασχόλησης ε, που κρέμονται από, ένα, από μια κλωστή γιατί οι επιχειρήσεις ε, ε κοιτούν μόνο το κέρδος τους, ε, τα κέρδη τους. Αλκόα, Vodafone, Deliveroo, Amazon, ένα, ένας τεράστιος κατάλογος, δεν χρειάζεται να σας το διαβάσω όλα. Αυτά είναι το αποτέλεσμα όταν αφήνουμε τη δημοκρατία στα χέρια των πολυεθνικών, όταν η προτεραιότητα είναι τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, όπου και αν βρίσκονται και από όπου και όταν προέρχονται. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε δημόσιε πολιτικέ που θα προωθούν τι ποιοτικέ θέσει απασχόληση και θα εμποδίζουν ναι, την εργασιακή εκμετάλλευση σε οποιαδήποτε από τα κράτη-μέλη, γιατί μέχρι τώρα η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων έχει προχωρήσει παράλληλα με την ελεύθερη κυκλοφορία τη φτώχεια και τη ανισότητα. Οι οικονομικέ πολιτικέ ε, ε, της, ε, ε, μην τις συνεχίζετε, μην προβαίνετε σε στήρε, σε Ε, επιτεθείτε στα προβλήματα που επηρεάζουν την εργατική τάξη. Δεν χρειαζόμαστε δεσμεύσει. Για παράδειγμα, ώστε η κοινωνική πολιτική να μετατραπεί σε ευρωπαϊκή πολιτική, να πιέσετε ώστε να επικυρωθεί ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Αυτό είναι ένα καλό κοινωνικό συμβόλαιο. Να κάνουμε την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική ένα παράγοντα σταθερότητα και όχι ε, και όχι αντιφάσεων όπως ας πούμε στην Δυτική Σαχάρα και στην Παλαιστίνη. Ε, ε, Εκλογικό νόμος, ε, ισότητα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, απειλείται η δεξιά, την έχουμε Δι, γυναίκες, στο, έχουμε ζήσει στο πετσί μας, είναι διαρθωτική, θα συνεχίσουμε ωστόσο να αγωνιζόμαστε για να περασπιστούμε τα κοινά μας συμφέροντα των γυναικών. Ευχαριστώ. Ελευθερία και Άμεση Δημοκρατία, η κυρία Φεράρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα μαζί μας εδώ. Πρόκειται για την 15η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης που γίνεται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για 15η φορά πρέπει να επαναλάβουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση διανύει μια πολύ δύσκολη στιγμή και για 15η φορά πρέπει να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο και η απάντησή μας είναι πάντοτε η ίδια. Λάθος πολιτικές, ε, αδικίες. Να σας δώσω μόνο δύο παραδείγματα. Οι πολιτικές λιτότητες έχουν προκαλέσει τεράστιες ζημιές στην κοινωνία μας. Εχθές ο πρόεδρος Γιούνκερ παραδέχτηκε σε αυτή την ολομέλεια ότι, ότι αυτές οι πολιτικές λιτότητες κάποιες ζημιές έχουν κάνει. Καλό, καλή αργά παρά ποτέ λέμε, αλλά εδώ όχι, έχουμε ήδη ξεπεράσει το, τα όρια. Έχουμε δημιουργήσει οικονομίες που έχουν διαλύσει το σύστημα προστασίας των εργαζομένων και των πιο ευάλωτων κατηγοριών, αφήνοντας ανικανοποιητές τις ανάγκες και... Ε, ε, Δημιουργώντα ανθρώπου που δουν σε δυσκολία, δράμα τη στόχιας, το δράμα τη έλλειψη απασχόληση και της κοινωνικός αποκλεισμός που ζουν εκατο, εκατομμύρια Ευρωπαίοι, δεν σημαίνει ότι είμαστε λαϊκιστέ. σημαίνει ότι διαπιστώνουμε την πραγματικότητα και προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσει. Ο Γιούνκερ και άλλοι επίτροποι εκμεταλλεύονται του τελευταίου μήνε που του μένουν στην Κομισιόν για τι επόμενε εκλογέ, θα υπάρξει αλλαγή μεγάλη, όχι μόνο στην Ολομέλεια, αλλά σε ολόκληρη την Επιτροπή. Το δεύτερο παράδειγμα που θέλω να αναφέρω στις λανθασμένες πολιτικές έχει να κάνει με τις μεταναστευτικές πολιτικές. Εδώ η αποτυχία της Ένωσης, μιας Ένωσης που είναι μόνο στα όνομα Ένωση και όχι στην πράξη, είναι προφανής. Η έλλειψη κοινή θέση για την ισότιμη κατανομή των ευθυνών και την αλληλεγγύη στις πολιτικές ασύλου και μετανάστευσης ανάμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη βήθησαν το μεταρρύθμιση ε, Τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, όσον αφορά το άσυλο. Αυτό σημαίνει πως ε, οι τα περισσότερα προβλήματα βαραίνουν τα συνοριακά κράτη κυρίως και τους λιγοστούς συνεργάτες τους. η αποτυχία αυτών των ευρωπαϊκών πολιτικών έχει μεγάλο αντίκτυπο και μεγάλο κοινωνικό κόστος και οικονομικό κόστος που εκτιμάται στα 49 ε, δις ευρώ, σύμφωνα με πρόσφατη ε, μελέτη. Δεν είναι η αλληλεγγύη μόνο που λείπει. Η Ισπανία και η Ιταλία είναι δύο χώρε τη Μεσογείου που έχουν τα ε, παρόμοια συμφέροντα, όπω α πούμε για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την οικονομία. Όμω, βλέπουμε την έκφραση δύο διαφορετικών πολιτικών δυνάμεων. Ωστόσο οι χώρες μας θα πρέπει να συνεργαστούν για να καταπολεμήσουν τα προβλήματα και να βρουν λύσεις για τα μεταναστευτικό. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να συμβάλλει. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να δώσουμε και άλλα μηνύματα στους πολίτες. Οι πολίτες μας ζητούν συγκεκριμένες δράσεις και απαντήσεις. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να περικόψουμε και τις ε, σπατάλες και ας ξεκινήσουμε από αυτήν εδώ, ε, αυτό εδώ το κοινοβούλιο, αυτή την άχρηστη και αδικαιολόγητη τριπλή έδρα. Ε, ε, ε, δισεκατομμύρια σπαταλώνται κάθε χρόνο για τα πηγενέλα. θα πρέπει λοιπόν να, να, καταργηθεί αυτή η σπατάλη. Αυτό δεν σημαίνει κατάρριση της δημοκρατίας. Η δημοκρατία δεν είναι, δεν είναι προνόμιο, ούτε ένα κτίριο μόνο. Η λιτότητα, τις σπατάλες, οι πολίτες μας ζητούν αλλαγές. Θα πρέπει οι άνθρωποι να μπουν στο επίκεντρο των πολιτικών και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να γίνει σεβαστό τώρα τα δικαιώματα και η ευημερία όλων των πολιτών και να μην θυσιάζονται στο όνομα συγκεκριμένων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ε, συμφερόντων που ευνοούν μόνο λίγους ανθρώπους. Ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, πριν από ένα χρόνο βρεθήκατε τυχαία στο επικεφαλής της Ισπανίας χάρη, λόγω του σκανδάλου που αντιμετώπισε ο Ραχώη. Ε, ωστόσο το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει μόνο 90 ε, έδρες. Είναι καταστροφικά τα αποτελέσματα για την Ισπανία. Η πρώτη σας κίνηση ήταν να δεχτείτε το Aquarius, ένα σκάφος το οποίο υποστηρίζει την παράνομη διακίνηση μεταναστών στην ε, Μεσόγειο, τη μαφία η οποία ε, πλουτίζει εκμεταλλευόμενη τις ανθρώπινες ζωέ. Οι διακινητές είναι αυτοί οι οποίοι υποφελούνται από την ε, διακίνηση αυτών των πλοίων όπου βάζουν τους μετανάστες. Ο Μακρόν και η Μέρκελ ε, ε, έσπευσαν να σας συγχαρούν. Ε, δεχθήκατε τις δύο, φορ... δύο φορές την κυρία Μέρκελ. Ε, χωρίς να διαβολευτείτε τους Ισπανούς, συνήψατε μία συμφωνία με την Καγκελάριο για να αντιμετωπίσετε το μεταναστευτικό. στο ζήλο σας δεν συνειδητοποίησατε ότι ε, μιλή, αναφέρθηκε στο Μαρόκο μιλώντας για μια αβυσαλαία ανισότητα. Ε, αυτή όμως είναι η πιο ευημερούσα χώρα ε, στην περιοχή. Μια συμφωνία επανεισδοχής είναι, θα ήταν πολύ πιο χρήσιμη. Ε, οι πρόσφυγες βέβαια μετά από την πολιτική που εφαρμόσατε έσπευσαν στις πόρτα σας. Ε, ε, στη Θέουτα και την ε, Μελίγια προσπαθώντας να παραβιάσουν τα σύνορα καμιά φορά και με τη βία. Είσαστε υποτελεί στο Βερολίνο αλλά και στις Βρυξέλλες. Το 2011 η σοσιαλιστική ομάδα έσπευσε να προβεί σε μια μεταρρύθμιση του Ισπανικού Συντάγματος όπου ε, η κυβέρνηση ε, ε, δεσμεύεται να δεχτεί τα όσα της βάλλονται από την Κομισιόν. Ωστόσο, ο Ισπανικός λαός πλέον αφυπνίζεται. Δείτε τι έγινε στην Ανδαλουσία και αναφέρομαι στο συνασπισμό κυβέρνησης που έδιωξε από αυτό το προπήγιο του σοσιαλισμού τους, ε, το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ε, το 2018 εξαιτία σας ε, η αύξηση των μεταναστών αυξήθηκε, ήταν δραματική. Στην Ιταλία, ωστόσο, το ποσοστό αυτό έπεσε σημαντικά γιατί οι Ιταλοί απέστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ε, διακινητές. Ο Ματέο Αλβίνη ε, δεν δέχεται ε, την εμπορία ανθρώπων η οποία αποφέρει περισσότερα κέρδη από το εμπόριο ναρκωτικών. Κύριε Πρωθυπουργέ, η επίλυση του μεταναστευτικού είναι συνάρτηση πολιτικής ε, βίλησης, βούλησης, γιατί ε, οι δικές σας ε, υπηρεσίες ακτοφυλακής είναι εξίσου αποτελεσματικές με τις αντίστοιχες ιτηλικές. Αλλά αντί να στηριχθείτε σε αυτούς, κάνετε προσπάθειες, δημιουργείτε ταμεία για την καλύτερη ένταξη των μεταναστών. parola all'onorevole non iscritto. Ο και μη Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό για τη δουλειά του, για την ε, ομιλία του. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, όταν έρχεται εδώ πέρα, δεν εκπροσωπεί το πολιτικό του κόμμα, αλλά εκπροσωπεί κυρίως τη χώρα του. Γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ την Ισπανία για όλες τις προσπάθειες της μέχρι στιγμής. Ακούσαμε τον συνάδελφο Φερχόφστατ που μίλησε για τον φεντεραλισμό. Η Ευρώπη σήμερα χρειάζεται πιο πρακτική προσέγγιση, περισσότερο σεβασμό για τις χώρες, ανταγωνιστικότητα ε, στην οικονομία και λιγότερο συγκεντρωτισμό. Αυτά ήθελα να ακούσω. Επίσης φαίνεται ότι έχουμε πολύ διαφορετικές απόψεις σχετικά με την αλληλεγγύη αλληλεγγύη είναι όταν βλέπω να υπάρχει ανάγκη να βοηθήσω κάποιον άλλον. Όταν κάποιος ε, έχει βρεθεί σε ατυχή θέση χωρίς ε, να ευθύνεται ο ίδιος. Δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να πληρώνω για την ανευθυνότητα των άλλων. Η Ισπανία θα είναι σημαντικός μας εταίρος κατά τη συζήτηση μιας πιο ρεαλιστικής προσέγγισης στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχει το λόγο ο κύριος ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους παρεμβαίνοντας και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό τον γύρο συζήτησης. Αν μου επιτρέπετε, ε, ε, θα ήθελα να πατήσω στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων από κοινού, όχι στον καθένα προσωπικά, γιατί αυτό θα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο. Η κεντρική ιδέα τη παρέμβασή μου είναι ότι θα πρέπει να προστατευτεί η Ευρώπη, ούτω ώστε η Ευρώπη να μα προστατεύσει και αυτή. Και πολλές από τις παρεμβάσεις των πολιτικών ομάδων έδειξαν ότι όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την Ευρώπη, ε, γευρώνοντας τις ε, πολιτικές μας διαφορές. Το ερώτημα είναι σε ποια κατεύθυνση και θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της μετανάστευσης. Ε, Βεβαίω ε, ισχύει τα ε, ε, δεν ισχύει το ότι η μετανάστευση ε, έφτασε μαζί με, το, με την άνοδο των σοσιαλιστών στην εξουσία. Αυτό το οποίο άλλαξε είναι η μεταναστευτική πολιτική στην Ισπανία, η οποία στο παρελθόν δεν είχε απολύτως κανένα νόημα. Εμείς πάντοτε ε, γνωρίσαμε τι γίνεται και αποφασίσαμε να δεχτούμε το Aquarius, γιατί γνωρίσαμε ότι η πρόκληση της μετανάστευση απαιτεί από όλες τις χώρες, από όλες τις χώρες ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια κοινή ε, θέση πρωτίστω το ανάληψη ευθύνη και δεύτερον την αλληλεγγύη. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ε, έχει μια εξωτερική ε, πολιτική όπως αυτή η οποία ανέπτυξε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Θα πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν βάσει των κονδυλίων να ενισχύσουμε την Αφρική. Εμείς εδώ ε, και μήνες έχουμε διμερείς ε, διαλόγους με το Μαρόκο και όλες τις χώρες του Σαχέλ, όχι μόνο ε, για τα συμφέροντα να προσπίσουμε τα της Ισπανίας, αλλά και ολοκλήρου της Ευρώπης. Η Ισπανία εδώ και πολλά χρόνια έχει μια πολιτική επιστροφής με το Μαρόκο, τη Μαυριτανία και άλλες χώρες της περιοχής. Εγώ πήγα στο Μαλί, όπου προσπαθήσαμε να, να επανεκκινήσουμε μια πολιτική εκούση ε, επιστροφής των υπηκών του Μαλή που αυτή τη στιγμή ζουν στην Ισπανία. Ε, προσπαθούμε να ενισχύσουμε λοιπόν αυτή την πολιτική επιστροφής ε, και προσπαθούμε επίσης να ενισχύσουμε την πολιτική στα σύνορα. Και χωρίς αμφιβολία αυτό που κάνουμε να ενισχύσουμε τις, ε, την πολιτική ένταξη. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να ενισχύσουμε αυτή την πολιτική ένταξη για όλους τους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και χωρίς αμφιβολία θα ήθελα να σας πω ότι είμαστε υπέρ μιας μεταρρύθμισης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χορήγησης Ασύλου. Ε, εμένα, εγώ εδώ έχω πολλές ανησυχίες όσον αφορά το Σέγγεν, γιατί υπάρχουν πολιτικές ομάδες όπως το ΕΛΚ που δεν συνεργάζονται εδώ. Με ανησυχεί λοιπόν η κατάσταση αυτή. Εμένα δεν με ανησυχεί τόσο πολύ η παρουσία της ακροδεξιάς. Αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι το πώς η ακροδεξιά παρισφρεί στην ατζέντα ε, πολιτικών κομμάτων που υποτίθεται ότι ήταν ε, φιλοευρωπαϊκά. Ε, η κυβέρνηση αυτή, κύριε Φέρχοφσατ, στηρίζει χωρίς αμφιβολία την έγκριση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Ε, το υπερασπιστήκαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και με την ε, προηγούμενη κυβέρνηση του κυρίου Ραχώη. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να εγκριθεί πριν από τις ευρωεκλογέ γιατί είναι θεμελιώδες για την ε, γεωργική πολιτική στην Ισπανία, πολιτική συνοχή και άλλες σημαντικές πολιτικές όπως είναι η πολιτική μετανάστευσης ή πολιτικές που συνδέονται με ζητήματα καινοτομίας. Εμείς ε, θα εγκρίνουμε τον ε, προϋπολογισμό της χώρας κατά πάσα πιθανότητα τον Απρίλιο. Ε, άρα λοιπόν αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται να προβούμε στην έγκριση του προϋπολογισμού γιατί θεωρούμε ότι είναι θετικός όσον αφορά την κοινωνική πολιτική και την αναδιανεμετική πολιτική και περιλαμβάνει καινοτομίες όσον αφορά το φορολογικό σύστημα, για παράδειγμα η δημιουργία φόρου επί των συναλλαγών και αυτά είναι κάποια από τα μέτρα που εσείς οι ίδιοι προτείνατε σε αυτό το σώμα και εμείς προωθούμε στο επίπεδο της εθνικής μας πολιτικής. Ε, επιτρέψατε μου επίσης να αναφερθώ για την Καταλωνία, γιατί ε, το έκανε η ε, επικεφαλή της πολιτικής ομάδας των Πρασίνων. Από το 2014 έγιναν πέντε ψηφοφορίες, ε, τρεις εκλογικές διαδικασίες σε περιφερειακό επίπεδο. Ε, ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτών των υποψηφισμάτων και αυτών των εκλογών ε, στο πλαίσιο του συνταγματικού ε, του Ισπανικού Συντάγματος. το 62% δεν υπερψήφισε την απόσχηση. Οι αποσχεσικές τάσεις δεν έχουν κοινωνική πλειοψηφία. Το 52% στην Ισπανία δεν είναι υπέρ της ε, απόσχησης. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να επιβληθεί ένα πολιτικό σχέδιο σε μια πλειοψηφία η οποία δεν συμμερίζεται την ε, απόσχηση. Πρώτο λόγο πρώτος λόγος είναι αυτός. Δεύτερον, είναι προφανές ότι στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Καταλωνία, εάν δούμε τι γίνεται για παράδειγμα στη Βαυαρία ή εάν δούμε τι γίνεται στο Βένετο στην Ιταλία ή στη Γαλλία, στην Κορσική, υπάρχουν εδαφικές ε, τάσεις, υπάρχουν ε, κινήματα εδαφικής ε, διάσπασης. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτό που συνέβη στην Καταλωνία και αυτό που συνέβη στο Βένετο ή για παράδειγμα στην ε, Βαβαρία όταν διάφοροι πολιτικοί σχηματισμοί ήθελαν να υπερσπιστούν την ανεξαρτησία της Βαβαρίας ή του Βένετο στην Ιταλία. Ή όταν το Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δικαστήριο του Βένετο στην Ιταλία ή ε, ε, αυτό που έγινε στη Βαβαρία. Στην ε, Ισπανία υπήρξαν κατ' επανάληψη αποφάσεις ε, του δικαστηρίου όπου υπόθηκε ότι δεν είναι δυνατή η απόσχηση. Ωστόσο, δεν εκπληρώθηκε αυτή η εντολή εκ μέρους των περιφερειών που επιθυμούν την απόσχηση. Από το 2010 η Καταλωνία έχει ένα σύνταγμα το οποίο στο σύνολό του δεν υπερψηφίστηκε από τους ε, πολίτες. Εδώ και δέκα χρόνια είναι προφανές ότι τα πολιτικά κόμματα όταν είναι στην αντιπολίτευση ε, χρησιμοποιούν ε, το θέμα της Καταλωνίας για να πιέσουν την κυβέρνηση. Ε, εμείς θα ακολουθήσουμε την πολιτική μας. Η Ισπανία είναι μια σημαντική χώρα η οποία έχει ένα υψηλό επίπεδο αποκέντρωσης, όχι μόνο οικονομικής αλλά και και πολιτιστική όσον αφορά την αναγνώριση των διαφορών γλωσσών και όσον αφορά τα παιδιά ε, που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν ένα εξαιρετικά υψηλό αίσθημα ε, εθνικό, ε, διαφορετικής, που έχουν διαφορετική εθνική προέλευση. Συγγνώμη. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι είναι προφανές ότι στην Καταλωνία θα πρέπει να γίνει μια ειλικρινής ε, διάλογος και να αναγνωρίσουμε ότι στην ε, Καταλωνία η πλειοψηφία δεν είναι εθνικιστική. Θα πρέπει να γίνει λοιπόν ένας διάλογος μεταξύ εθνικής κυβέρνησης και Καταλωνίας όσον αφορά την εθνικιστική, το εθνικιστικό και μη εθνικιστικό κομμάτι στην ε, Καταλωνία. Και βεβαίως ε, σημαντικό είναι το να έχει η ισπανική κυβέρνηση την πολιτική βούληση να επιλύσει το ζήτημα της Καταλωνίας. Αλλά θα πρέπει, όπως είπα, να αναγνωρίσουμε ότι οι αποσχετικές τάσεις δεν έχουν την πλειοψηφία στην Καταλωνία. Και ε, θέλει η κοινωνία της Καταλωνίας επιθυμεί μία λύση για, να, για το πρόβλημα αυτό. Η λύση που θεωρώ ότι υπάρχει στο ζήτημα των μεσοσυχών τάσεων είναι η βούληση να υπάρξει δυνατότητα συνύπαρξης. Τέλος, ο κ. Βέμπερα έκανε μια αναφορά στην πρόταση μορφής. Η πρόταση Μομφής είχε μια εντολή δηλαδή η δημοκρατική αναγέννηση της χώρας μας. Αυτό που συνέβη στην Ανδαλουσία, ανάμεσα στο ε, Λαϊκό Κόμμα, τους φιλελεύθερους και τους ε, αδερφούς του, ε, του Εθνικού Μετώπου της Γαλλίας, είναι μία ε, συνεργασία των δικαιωμάτων, μια συγχώνευση των δικαιωμάτων, όπως ας πούμε για την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση της ε, έμφυλης βίας. Στην Ανδαλουσία λοιπόν πέρασε ένα σύνορο το οποίο υπάρχει στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να κάνει συμμαχία με την άκρα δεξιά. Ποτέ δεν πρόκειται εμείς να το κάνουμε αυτό ε, όπως κάποιοι είπαν με τις θέσεις τους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να σας πω ότι η θέση της Ισπανικής κυβέρνησης είναι υπέρ της Ευρώπης. Αυτές είναι οι προτάσεις που είχαμε να κάνουμε. Τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων, τη στρατηγική ή μάλλον καλύτερα την καταπολέμηση της επισφάλειας στην εργασία την ε, ανεργία των νέων, ε, όλα αυτά τα πράγματα που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της Ευρώπης ώστε να μας προστατεύσει καλύτερα, ιδιαίτερα να προστατεύσει τους πιο ευάλωτους. Σίγουρα στην, Ευρωπαϊκή, στην Ισπανική κυβέρνηση και το Ισπανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα θα βρουν σύμμαχο. Κύριε Φερχόφσας, να σας πω και κάτι ακόμα. Ξέρετε πως... ε, ε Εσεί είστε πολλά χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο και εγώ μόλι 7 μήνε στην κυβέρνηση τη Ισπανία και σίγουρα μπορούμε να συζητήσουμε τα προβλήματά μα. Όμω, πιστεύω πω θα πρέπει να βρούμε και εξόδου σε αυτό το, την έλλειψη ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων που χρειάζονται στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη εξωτερική Πολιτική. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αλλαγή των διαδικασιών λήψη απόφαση στο Συμβούλιο και στο, στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν. Και σίγουρα, όπω το είπα ήδη, θα προσπαθήσουμε να αλλάξουν ε, οι κανόνες ώστε να μην λαμβάνονται αποφάσεις ομόφωνα μόνο. Όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, θα χρειαστεί βέβαια αλλαγή στις συνθήκες, για άλλα πράγματα όχι. Ο Υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Μπορέλ, μόλι μου θύμωσε, θύμισε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τι πασαρέλε που υπάρχουν ε, στι συνθήκε για να ενισχύσουμε τον γενικό χαρακτήρα της Υπήρου μας ε, στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινάμε με τον Catch the Eye. Καθυστερούμε λίγο τις ψηφοφορίες σας. Παρακαλώ να σεβαστείτε το ένα λεπτό, γιατί όσο περισσότερο το σεβαστείτε, τόσο περισσότερο θα πάρετε και το λόγο. 150 έχουν ζητήσει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ζούμε σε μια εποχή ψευδών ειδήσεων, αλλά επίσης και όπως είδαμε και σε μια εποχή ε, σφαλμένων και ψευδών επεπιθύσεων. Με, την ψήφο των, ε, πρώην τρομοκρατών και της άκρο αριστεράς βρίσκονται στην εξουσία αυτή η κυβέρνηση. Και μόνο με τις ψήφους των αποσχιστών, των πρώην τρομοκρατών και της ακροαριστεράς θα μπορούσαν να σταθούν. Οι πρώτη σας ομιλίες μιλήσατε πολύ για την παγκοσμιοποίηση, αλλά δεν μπορέσατε να μιλήσετε για την ενότητα της Ισπανίας και δεν μπορέσατε να υπερασπιστείτε το κράτος δικαίου. Μιλήσατε, θα σας πω κάτι για την Καταλωνία. Αυτό που είπατε είναι, είναι ότι δεν είναι πρόβλημα ανεξαρτησίας, αλλά πρόβλημα συμβίωσης. Ενώ το ανώτατο δικαστήριο α, ξεκινά τέτοια διαδικασία και όλοι περιμέναμε τον πρόεδρο της Ισπανικής Κυβέρνησης να υπερασπιστεί το κράτος δικαίου της χώρας μας. Και το λέω ως Ισπανός βουλευτής. Δύο χρόνια υπερασπιζόμαστε και τους δικούς σας βουλευτές εδώ για την ενότητα της Ισπανίας. Αλλά το να υπερασπιστείτε την ενότητα της Ισπανίας είναι μόνο θέμα της θέσης σας, αλλά είναι και θέμα πεποίθησης, πε, που να μην είναι ψευδής. Δυστυχώς, επειδή είστε πρόεδρος της Ισπανίας στην, στην Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν σας βγήκε εσείς, εσ, εσείς δυστυχώς δεν μπορέσετε να το κάνετε. Με, με αλλά κάνω υπομονή. Κυρία Γκαρσία Πέρες, Πρόεδρε Σάντσες. Είναι ευαίσθητη, λεπτή στιγμή για την Ευρώπη. Και το να ακούμε την ομιλία σας με δέσμευση σαφή για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ανανάσα για όσους πιστεύουμε ότι η λύση στα προβλήματά μας βρίσκεται στην Ευρώπη, σε περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Δεν μπορούμε λοιπόν να αντισταθούμε στον πειρασμό να φέρουμε αυτά τα επιχειρήματα στη Μαδρίτη για να κερδίσουμε, να, να μην διστάσετε μάλλον να τα φέρετε στη Μαδρίτη για να κερδίσετε πόντους αλλά δεν θα εξυπηρετήσουμε την Ευρώπη αν δεν χρησιμοποιήσουμε αυτό το χώρο και την καρδιά της Ευρώπης για να μιλήσουμε για το πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου. Περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, περισσότερη ισορροπία, να αποφύγουμε τις ανισότητες, να προωθήσουμε μια Ευρώπη όπου να υπάρχει ισότητα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, να μπορούμε να κοιτάξουμε στο καταπρόσωπο πρόσωπο τους, τους πολίτες και να πούμε πως η Ευρώπη είναι τη λύση για τα προβλήματα. Αυτή είναι η δέσμευση των Ευρωπαϊστών, της σοσιαλδημοκρατίας και θα πρέπει να, να δουλέψουμε και να προσπαθήσουμε με νύχια και με δόντια ώστε να υπερασπιστούμε περισσότερη Ευρώπη που θα μπορεί, όπως είπα, να κοιτάξει κατά πρόσωπο τους πολίτες. Και ευχαριστώ πολύ που μπορείτε να έχουμε να έχουμε κυβερνήσεις ε, μέσα στην Ευρώπη που, θα εξακολουθούν να στηρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Η πολιτική ξεκινάει με την παρατήρηση της πραγματικότητας, έχει πει ένας ε, γνωστός ε, σοσιαλδημοκράτης ε, και γι' αυτό γιορτάσαμε την επέτειο του ευρώ και άκουσα έξι ομιλίες που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μάλλον επιθυμίες εξέφρασαν. Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλετε κοινωνική Ευρώπη. Η κοινωνική Ευρώπη δίνει δουλειά στους ε, πολίτες και προοπτικές στους νέους. Αυτό είναι αποφασιστική σημασίας. Θα πρέπει λοιπόν να ρωτήσουμε γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη ανεργία στους νέους, ε, γιατί δεν ε, έχουμε ιδιωτικές επενδύσεις, ε, υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα στην Ευρώπη. Υπάρχουν επισφαλείς θέσεις εργασίας σε άλλες χώρες. Εργαζόμαστε όλο και περισσότερο για λιγότερα χρήματα και δεν είναι αυτή η κοινωνική Ευρώπη που θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ. Αντιμετωπίζουμε την απειλή των λαϊκιστών και αποσχιστών. Αλλά δεν αρκεί η καταγγελία. Θα πρέπει να δώσουμε αποτελεσματικές απαντήσεις στην αιτία που είναι η αλλαγή μοντέλου η σύγχυση που επικρατεί στην οικονομία. Ωστόσο σήμερα όλο έχουμε δόγματα παρά λύσεις. Κύριε Σάντσεθ, η λύση δεν είναι με τους λαϊκιστές της αριστεράς ή της δεξιάς που θέλουν να αποδυναμώσουν την Ευρώπη ενώπιον του λαϊκισμού και της απόσχεσης των αποσχιστικών τάσεων θα πρέπει να προσπαθήσουμε να οικοδημήσουμε την Ευρώπη και να την υπερασπιστούμε. Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω σε εκείνους που θεωρούν ότι η Καταλωνία είναι πρόβλημα των Καταλανών, ότι στην Καταλωνία το πρώτο κόμμα το οποίο αναπτύσσεται στην Ισπανία είναι το κόμμα Σιουδαδάνος, όχι κόμμα αυτονομιστών. Αρκεί τον, φτάνει, δεν χρειάζεται να προβάλλουμε άλλα συνθήματα. Ε, βασική μας αρχή θα πρέπει να είναι η ελεγγύη και η ενότητα. Αυτό ισχύει τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ισπανία. Κύριε πρόεδρε της Ισπανικής Κυβέρνησης στις 5 Νοεμβρίου του περασμένου έτους ε, πήγα να επισκεφτώ τους παλιούς συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που σήμερα είναι φυλακισμένοι στις Ισπανικές φυλακές. Ε, κάτι που σήμερα ε, είναι αδιανόητο να βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Άνθρωποι οι οποίοι εξελέγησαν καταρχήν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη συνέχεια στην Καταλωνία με νόμιμο τρόπο να φλαγίζονται για τις ε, πολιτικές τους ιδέες. Έχουμε στο Κοινοβούλιο αυτό κατ' επανάληψη πει και καταγγείλει τις ανελεύθερες ε, πολιτικές του κυρίου Ορμπάν. Έχουμε καταγγείλει την ανελεύθερη πολιτική της Πολωνίας Έχουμε καταγγείλει απολύτως δικαιολογημένα τις επιθέσεις στα δικαιώματα που σήμερα λαμβάνουν χώρα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα λοιπόν η Ισπανία λόγω ακριβώς του συντάγματός της και της πολιτικής η οποία εφαρμόζεται στην Καταλωνία προσχωρεί στο στρατόπεδο αυτών των χωρών. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι κρίμα. Άκουσα την ομιλία σας. Αλλά πώς είναι δυνατόν ε, σήμερα ε, άτομα, βουλευτές συγκεκριμένα, μέλη περιφερειακών κυβερνήσεων ε, και ενώσαν να είναι φυλακισμένοι. Άκουσα την έκκλησή σας για το διάλογο και τη συμμερίζομαι αλλά θα πρέπει να απελευθερώσετε άμεσα αυτά τα άτομα προκειμένου να υπάρξει διάλογος. Ε, θα πρέπει να αναλάβετε τις ε, ευθύνε σας. Ε, απελευθερώστε άμεσα τα άτομα αυτά, μόνο έτσι θα αποδείξετε το δημοκρατικό σας πνεύμα. Ε, Πρώτα, σας υπενθυμίζω ότι πρέπει να σεβαστούμε το σύστημα DONT. Εάν δεν τηρήσετε το χρόνο αγόρευσης, ε, αυτό θα είναι σε βάρος ενός συναδέλφου. Αυτό είναι ο κανόνας και θα πρέπει να την, ε, το σεβαστείτε. Ο κύριος Ορμπαν Κρέσπο. Κύριε Σάντζε, η κυβέρνησή σα ξεκίνησε υποδεχόμενη το Aquarius και έξι μήνε αργότερα τελείωσε μπλοκάροντας το Open Arms στη Βαρκελόνη και σίγουρα προς χαρά φασιστών όπως ο Σαλβίνη. Υποσχεθήκατε την εξαίρεση ε, και την άρση του νόμου Φήμοτρο, αλλά συνεχίζει να ισχύει. Υποσχεθήκατε την ε, εργασιακή μεταρρύθμιση. Όχι μόνο θα το κάνατε, αλλά επιτρέψετε και σε εταιρείε όπως η Αλκοά να απολύουν ε, εκατοντάδες εργαζόμενους. Υποσχεθήκατε φόρο στις τράπεζες ε, αλλά δεν έχει φτάσει. Υποσχεθήκατε να ρυθμίσετε τη φούσκα των ε, ε, μισθωμάτων που, που διώχνουν από τα σπίτια τους εκατοντάδες ανθρώπους, αλλά τίποτα δεν κάνατε. Τελικά κερδίζουν τα αρπακτικά νεοφιλελεύθερες πολιτικές σε αυτές τις ένοχοι, στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της ε, Μεγάλης Συμμαχίας και στην Ανδαλουσία χρειαζόμαστε ε, μία στροφή 180 μοιρών από τις πολιτικές περικοπών που εξυπηρετούν τις ελίτ. Είναι σημαντικό να γίνει αλλαγή στην Ευρώπη. Δεν έχουμε πια χρόνο κύριε Σάντσες, πρέπει να γίνει τώρα η αλλαγή. Ο κύριος Ντάρμος. Ε, Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κύριος Μποβέ σχετικά με τους Καταλανούς φυλακισμένους ε, που επί ένα χρόνο κρατώνταν πριν τη δίκη τους. Πρόκειται για πολιτικούς κρατούμενους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως δεν κάνει τίποτα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν κάνει τίποτα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο δεν λέει τίποτα. Και ακόμη και ο κύριος Φερχόφστατ σιωπά. Οι ευρωπαϊκές αξίες για τις οποίες ακούμε συνέχεια ε, δεν γίνονται σεβαστές και αναρωτιέται κανείς γιατί η Ισπανική κυβέρνηση στηρίζει το ευρωπαϊκό εγχείρημα και γι' αυτό φαίνεται ότι είναι εντάξει το να έχει κανείς πολιτικούς κρατούμενους. Αυτό είναι λυπηρό. Η υποκρισία είναι πολύ δύσκολο να παταχθεί και καλό όλους σας να κοιταχτείτε στον καθρέφτη και να αρχίσετε εκστρατεία για απελευθέρωση αυτών των πολιτικών κρατούμενων. Ο κύριος Καλώ ήρθατε κύριε Πρωθυπουργέ. Έχω κάποια ερωτήματα να σας ε, υποβάλω. Ποια πρακτικά, σε, ποιε πρακτικέ ποιες πρακτικές ενέργειες θα προβείτε ούτως ώστε η χώρα σας, η Ισπανία, η Ιταλία αλλά και η πατρίδα μου Ελλάδα να πάψουν να είναι τόποι μόνιμης διαμονής παρανόμων μεταναστών. Είπατε ότι είστε υπέρ της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Στρατού. Για να δικαιολογείται όμως η αύξηση των δυνατοτήτων των στρατιωτικών της ευρωπαϊκής ενώσεως θα πρέπει να υπάρχει ένας εχθρός ο οποίος θα απειλεί την ευρώπη. μπορείτε να μας κατονομάσετε ποιος είναι αυτός ο εχθρός και ποιες χώρες απειλεί διότι όπως ξέρετε και όπως γνωρίζω και εγώ οι μόνες χώρες της ευρώπης που απειλούνται από τρίτη χώρα είναι η ελλάδα και η κύπρος που απειλούνται από την τουρκία. είπατε επίσης ότι η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει έξω από τα σύνορά τη. αυτή είναι η ευρώπη του μέλλοντος που τότε θα μειωθεί η δύναμη των κρατών και κυρίως των μικρών κρατών. μπορείτε να φανταστείτε τη χώρα σας να θίγεται να θίγονται τα συμφέροντά της να βρίσκεται στην θέση της μειοψηφίας και να μην μπορεί να υπερασπιστεί αυτά τα συμφέροντά της. ευχαριστώ. Yes, thank uh, σας ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ. Καταρχάς για μια πολύ επικοδομητική ομιλία. Είναι σαφές ότι η ε, Ισπανία είναι αξιόπιστος ετέρος της Ευρώπη και η Ευρώπη είναι αξιόπιστος εταίρο της Ισπανίας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν ε, την πολιτική συνοχή σε την εγγύηση για τους νέους. Ας είμαστε σαφείς όμως, η ευθύνη για μια κοινωνική Ευρώπη ξεκινάει στα σπίτια μας, ε, στις πατρίδες μας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι επικίνδυνη στρατηγική ε, να ε, ρίχνετε στην Ευρώπη το φταίξιμο για αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς ε, στη χώρα σας. Η Ισπανία βρίσκεται σε καλή θέση λόγω της καλής δουλειάς προηγούμενων κυβερνήσεων. Να συνεχίσουμε λοιπόν αυτή την εργασία και ας μην ρίξουμε σε επόμενες γενιές τον φόρτο προσβλέπω στη συνέχιση τη συνεργασία με την Ισπανία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λόπες Ιστουρίς. Κύριε Σάντζες. Σήμερα εδώ μιλάμε για το μέλλον της Ευρώπης και δεν κατάλαβα γιατί τελικά η ομιλία σας ε, μετατράπηκε σε μια μικρή προεκλογική ομιλία υπέρ του κυρίου Τίπερμανς, ε, Τίμερμανς. Και επίσης αναρωτιέμαι γιατί αυτοί που χρησιμοποιούν τους ε, παλιούς δικτάτορες για να καταδικάσουν άλλους γιατί δεν μιλάτε για τους σημερινούς δικτάτορες όπως της Βενεζουέλας και της Κούβας. Εσείς θα ζητήσετε ε, κυρώσεις εναντίον αυτών των δύο ή θα συνεχίσετε μόνο με λόγια. Θα δείξετε τον φιλοευρωπαϊσμό σας καταγγέλλοντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μη στηρίζοντα τα δικτατορικά καθεστώτα του Μπαντούρο και του Κάστρο γιατί ο Κάστρο είναι που ε, που ηγείται της Κούβας. Ε, υπάρχουν ε, πολιτικοί κρατούμενοι στην Κούβα και στη Βενεζουέλα και τότε θα πούμε και εμείς ότι είστε ευρωπαϊστής. Μπλάνκο Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Στέμπαν Γκοσάλε Πόνσο, το να είναι κανείς πατριώτης ε, δεν σημαίνει το να στηρίζει την Ισπανία, αλλά να τηρεί τις συνταγματικές και ευρωπαϊκές αρχές και όχι να ε, πάει χέρι-χέρι με αυτόν που θέλει να τις καταστρέψει. Εσείς είχατε την ευκαιρία να δείξετε ότι είστε πατριώτης Ισπανι... Ισπανός, στηρίζοντας την κυβέρνηση της Ισπανίας, όπως ανέκαθεν κάναμε εμείς οι σιωλισσαλιστές, όταν η Ισπανία το και εσείς ερχόσασταν να μας ζητήσετε βοήθεια. Εσείς όμως στάσατε στην κυβέρνηση Τη Ισπανίας φωνάζοντας θα διαλυθεί η Ισπανία ενώ τούτη η Ισπανία ε, έλαβε μια Ισπανία με σε μια Ισπανία πιο διχασμένη από ποτέ με συνύπαρξη και συμβίωση ε, χειρότερη από ποτέ. Δυστυχώς εσείς δεν συμβάλλετε στο να δημιουργηθούν χώροι συμβίωσης που είναι ακριβώς αυτό το οποίο στηρίζει η κυβέρνηση της Ισπανίας η σημερινή. Και ευχαριστώ. Ο κύριος Τόμασιτς. Σα σας ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε κύριε πρωθυπουργέ σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας στη συζήτηση αυτή μετά το δημοψήφισμα για το Brexit και με την εκλογή του Προέδρου Τραμπ ε, ε, κινούμαστε προς ε, μια πολύ κακή κατεύθυνση. Εσείς αναφερθήκατε σε σημαντικές προκλήσεις που δεν ε, σχετίζονται με την πολιτική ολοκλήρωση όπως είναι τα εργασιακά δικαιώματα και θέματα της κοινωνικής Ευρώπης. Η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει να είναι προπίδιο των ε, εργασιακών δικαιωμάτων για να είμαστε όμως ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο δεν θα πρέπει να εισάγουμε αδικαιολόγητα υψηλούς φόρους και ε, αυστηρή, υπερβολικά αυστηρή νομοθεσία. Το θέμα αυτό σχετίζεται και με τις δημόσιες δαπάνες. Επί πολύ καιρό η Ισπανία αντιμετώπιζε προβλήματα ή ε, θα είναι σημαντική όμως για το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ, Κύριε Πρωθυπουργέ, ε, αναμένουμε να ε, φέρετε ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο να οικοδομείται με εμπιστοσύνη. Ε, εμείς η χώρα των Βάσκων θέλουμε να συμβάλλουμε στη σταθερότητα, να συμβάλλουμε σε μια χώρα που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις, ενισχύει το σύστημα κοινωνικής προστασίας ε, προωθεί εγχειρήματα τα οποία επιφέρουν ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Ενώπιον σύνθετων προβλημάτων χαιρετίζουμε τη βούλησή σας να τα επιλύσετε. Ε, ωστόσο, ε, πουλάτε... Δεν θέλουμε να πουλήσετε εσφαλμένες συνταγές. Ε, θέλουμε να υπάρξει ένα μοντέλο συνύπαρξης, το οποίο όμως να εδράζεται στον νόμο. Δεν είναι δυνατόν να μετατραπεί ένα πολιτικό πρόβλημα σε μια νομική υπόθεση. Ε, θα πρέπει να υπολογίστε στη δική μας ε, συνεργασία εάν θέλετε να επιφέρετε αποτελέσματα χρήσιμα και υποφελή για τη συνύπαρξη, την ελληνική συνύπαρξη όλων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σάντσεφ, ε, χαιρετίζουμε την ε, παρουσίαση του προπολογισμού στην Ισπανία γιατί ε, μας υπενθυμίζετε ότι είναι δυνατόν στην Ευρώπη ένας πιο σοσιαλιστικός κοινωνικός ε, δρόμος. Ε, απέναντι στην Ευρώπη του μίσους υπάρχει και το μοντέλο της βιώσιμης Ευρώπης. ένα μοντέλο πιο φιλόδοξο όσον αφορά την επίδειξη τόλμης έναντι του μεταναστευτικού ε, εφόσον επιτρέπεται την υποδοχή σκαφών που σώζουν ζωές και βαίνουμε προς, μια, ε, προς τη μετάβαση ενός πιο οικολογικού μοντέλου. Ε, είστε υπέρ των καθαρών συνεργειών, υπέρ της κλιματικής προστασίας, υπέρ της μείωσης των, της ρήπανσης του περιβάλλοντος. Όλα αυτά βρίσκονται στα χέρια σας. Θα σας στηρίξουμε. Ο κύριος Κόμη. Καλημέρα σα, ε, Πρόεδρε. Καλώ ορίσατε ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εσεί μιλήσατε πολύ για τι γυναίκε, για τα δικαιώματα των γυναικών, τη βία κατά των γυναικών. Εύχομαι την επόμενη φορά να μπορέσετε να μα έρθετε με κάπω πιο θηλυκό επιτελείο, γιατί σήμερα μόνο άνδρες βλέπω. Από τα λόγια να περάσουμε στι πράξει. Ε, ε, αυτή είναι η ευχή μου λοιπόν. Τώρα επειδή η Ιταλία και η Ισπανία ανέκαθεν είχαν καλή σχέση και, ξεκινώ, για την μετανάστευση πιστεύω πως ε, εκεί μπορούμε να είμαστε οι εκπρόσωποι των χωρών της, της Μεσογείου για τη μεταρρύθμιση της, μεταρρύθμιση της του Δουβλίνου. Και γιατί όταν λέμε ότι πως η Ευρώπη μας άφησε μόνος, ε, υπάρχει όνομα και επίθετο. Είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπάρχουν τα κράτη-μέλη. Τα Ευρωκοινοβούλια υποψήφισε τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου και τις ε, ε μεταναστευτικέ Όμως Όμω εσεί και οι άλλοι πρωθυπουργοί θα πρέπει να συμφωνήσετε για το θέμα για τις βίες κατά των γυναικών. Εμεί στο ΕΛΚ είμαστε υπέρ να υπάρξει ένας απολογισμός, ένας ε, σύνδεσμος που μπορεί να είναι αυτός των, ε, ε, της απασχόλησης και της οικογένειας και οι γυναίκες να μπορούν να εργάζονται και να μην κάνουν μόνο τις νοικοκυρές υποχρεωτικά και όχι από επιλογή. Ο κύριος Φέρμπερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρωθυπουργέ όταν συγκρίνεται την Καταλωνία και τη Βαβαρία. Θα ήθελα να ε, δίδεται ακριβή στοιχεία. Ε, πριν από 100 χρόνια υπήρξε μια ακροαριστερή ε, κίνηση για απελευθέρωση σε μια εποχή που δεν υπήρχε το βασίλειο της Γερμανίας. δεν είναι συγκρίσιμη με την περίπτωση της Καταλωνίας η περίπτωση αυτή. Δεύτερον, ε, είπατε τι θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό ε, επίπεδο. Εγώ θα ήθελα να ακούσω και τι κάνει η κυβέρνησή σας. Ε, δεν αρκεί να απαιτείτε λύση στην ανεργία από πλευρά της Ευρώπης τη στιγμή που ανακαλείται με τα ρυθμίσει της προηγούμενης κυβέρνησης για απελευθέρωση της αγοράς εργασίας. Εσείς δηλαδή δεν λαμβάνετε μέτρα για την απασχόληση των νέων. Ε, ήθελα να ακούσω περισσότερα για το θέμα αυτό. Δεν αρκεί να ζητάτε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Θα πρέπει κανείς να λαμβάνει και μόνος του μέτρα. Ε, είναι θέματα αλληλένδετα μεταξύ τους αυτά τα πράγματα. Παρακαλώ. Köszönöm Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε εδώ για το μέλλον της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Σύστημα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Υπάρχουν ε, κυβερνήσεις κρατών μελών ε, που ε, δεν δέχονται ανθρώπινα δικαιώματα και δημιουργούν ένα σύστημα ε, μη φιλελεύθερο και αναφέρομαι στην Ουγγαρία και ε, τον Βίκτορ Ορμπάν. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, έχουν αλλάξει και οι βουλευτές δεν κάνουν τίποτα. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν αποκτήσει τεράστιες περιουσίες, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες παιδιών πεινούν. Επίσης ε, παρενοχλούνται ε, άνθρωποι ε, της κοινωνίας των πολιτών. Η Ισπανία από δικτατορία έχει γίνει μια σεβαστή δημοκρατική χώρα. Τι πρέπει να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφύγουμε τις δικτατορίες στο μέλλον. Ευχαριστώ. Αν μιλάτε το διπλάσιο από το χρόνο που σα έχει δοθεί, παίρνετε το χρόνο των συναδέλφων σας. Στη μία η ώρα θα ψηφίσουμε. Καλώ ορίσατε κύριε Σάντσε, ε, κύριε Δεμεσμάκερ. Στις 21 ε, Δεκεμβρίου ήμουν στη Βαρκελόνη και εσείς ήσασταν εκεί. Ε, τέσσερις Καταλανοί κρατούμενοι είχαν μόλις σταματήσει την απεργία πείνας. Εγώ δεν ε, μου πέφτει λόγος για τις πολιτικές σας και τις στρατηγικές σας. Αυτό που δεν δέχομαι όμως είναι ότι ο κόσμος τώρα εδώ και πάνω από χρόνο βρίσκεται στη φυλακή λόγω και κατηγορούνται για ε, απόσχηση. Κανένας δεν έχει κάνει ε, βίαιη ε, επανάσταση και δεν το βλέπουμε αυτό σε ε, χώρες όπως η δική μου. Οι πολιτικές επιδιώξεις στηρίζονται μέσω του, διαλόγου. Νομίζω πως έχετε χάσει εδώ μια στιγμή. Υπάρχει, αυτή, υπάρχει επικίνδυνη εθνικισμός στην Καταλωνία ε, όχι όμως στην Καταλωνία, με συγχωρείτε, αλλά ε, αλλού όπου αναβιώνει ο φραγκισμός και ελπίζω πως θα ξεπεράσετε το φόβο σας ε, των άκρων και θα απελευθερώσετε τους πολιτικούς κρατούμενους. Ο κύριος Τρεμόζα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ Σάντσες, Κύριε Μπορέλ, καλώς ήρθατε και πάλι στο Ευρωκοινοβούλιο. Ε, δημιουργήθηκε ένα φοβερό προηγούμενο στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί φυλακίσατε τους καταλανούς ηγέτες πέρυσι. Πιο καλά στην Τουρκία είμαστε, στην Ισπανία και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να γίνει ρεφερέντουμ, δημοψήφισμα που δεν είναι έγκλημα για τη μεταρρύθμιση του Θαπατέρου από το 2005. Επίσης, κανονικά ε, υποτίθεται ότι τα καταλανικά είναι επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο φεντεραλισμός είναι να μπορούμε να μιλάμε τη γλώσσα του άλλου. Ποια μέρα θα μιλήσουμε καταλανικά εδώ μέσα και έπειτα. Στην Καταλωνία δεν έχουμε πρόβλημα συμβίωσης. Το πρόβλημα είναι η κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας. Ε, στο διάλογο θα τα βρούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. μου κύριε Πρόεδρε να ξεκινήσω λέγοντας ε, ότι ε, αφού αναφέρεστε για τον εξτρεμισμό το πρόβλημα είναι ότι στην πραγματικότητα δεν ε, εφαρμόζεται τίποτα από τις αρχές σας. Αυτή τη στιγμή ε, μια πρόταση εμπιστοσύνης τελικά τερμάτισε τη θητεία του Ραχώη. Εσείς πέσατε στην αγκαλιά των πολιτικών κομμάτων των αποσχιστών οι οποίοι προσπάθησαν να διαρρήξουν τη συνταγματική τάξη, οι οποίοι παρεκτράπηκαν από τον νόμο και δεν έχουν καμία δημοκρατική νομιμότητα. Κύριε Πρωθυπουργέ, μπορείτε να έρθετε εδώ και να μας αφηγείτε μια ιστορία, αλλά όταν στο τέλος η πραγματικότητα και τα δεδομένα τελικά αποκλίνουν τόσο πολύ, θα συνειδητοποιήσετε τι γίνεται. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια και εσείς δεν έχετε καμία απολύτως συνέπεια και το αποδείξατε. Κύριε κύριε Πρωθυπουργέ, Αναφερθήκατε στη νέα νομιμοποίηση της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Ζητήσατε περισσότερη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Δεν πιστεύετε ότι οι πολίτες ε, βρίσκουν ότι έχουν στερηθεί την κυριαρχία τους, ε, δεν μπορούν πια να αποφασίσουν για το ίδιο το μέλλον τους. Βλέπουμε από βιομηχανοποίηση ε, και εγκατάλειψη πολλών περιοχών και οι άνθρωποι που μένουν εκεί ε, θεωρούν ότι δεν έχουν ελέγγυν ως προς το πώς ε, θα εξελιχθεί η ζωή τους. Πώς βλέπετε εσείς την κυρίαρχη δημοκρατία η οποία με νέο τρόπο θα αντιστοιχεί στην επιθυμία των πολιτών να έχουν λέγει όσον αφορά το μέλλον τους. Όλα αυτά ε, σε συνδυασμό με την ιδέα ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο ξεκίνημα. Αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ, ήταν κεντρικό σε όλα τα θέματα που συζητήθηκαν από το Brexit μέχρι την Καταλωνία. Ευχαριστώ, Σαλαφράγκα. Κύριε Πρόεδρε τη Κυβέρνηση, καλώ ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το είπατε με βεβαιότητα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε αξίε. Γι' αυτό αυτό το Κοινοβούλιο έχει ε, ε, μια παρέγκλητη δέσμευση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει σε οποιαδήποτε χώρα ή ήπειρο. Ε, είναι καθολικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό και φτιάξαμε αυτό το βραβείο για την ελεύθερη ε, συνείδηση που ονομάζεται Ζαχάροφ. τρία, έχουμε δώσει μάλλον ε, στον Οσβέλτο Βάνια, τον Γουλιέλμο Φαρίνια και πέρσι στην δημοκρατική αντιπολίτευση της ε, τα βραβεία Ζαχάροφ. Εσείς τι άποψη έχετε. Πιστεύετε ότι οι βραβευμένοι είναι αξιόλογα άνθρωπα, τα ε, άτομα τα οποία υπερασπίζουν την ελευθερία και την αξιοπρέπειά τους, είτε είναι στην Κούβα είτε είναι στη Βενεζουέλα. Θα είσαστε διαθέσιμος να συναντηθείτε μαζί τους και σε σχέση με τη Βενεζουέλα έχουμε ε, με μεγάλη πλειοψηφία ε, ψηφίσει ψήφισμα που ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να ε, ζητήσουν ε, ε, να γίνει έρευνα από το, Ευρωπα... από το Διεθνές Δικαστήριο για τα εγκλήματα που έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα. Και ποια είναι η γνώμη σας αν ζητήσουμε από τον Καναδά και τις είπα να συμφωνήσουν για αυτή τη διαδικασία. κυρία Βαλενσιάνο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, εσείς σκεφτήκατε ότι το ο ΕΛΚ ε, που έχασε την πλειοψηφία. Όχι. Ε, το ΕΛΚ ζητάει ένα πατριωτισμό όταν είναι στην αντιπολίτευση αλλά οι ίδιοι από την πλευρά τους δεν ε, το κάνουν όταν εμείς είμαστε στην κυβέρνηση. Η βασική ιδέα που διαβιβάσατε εδώ είναι ότι πνέει ένας αέρας λαϊκισμού ε, κατάτμισης, διέρεσης, εξτρεμισμού στην Ευρώπη, ε, αντιδραστικού πνεύματος έναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έναντι στην ισχύ της Ένωσης, έναντι στην ε, ε, ισχύ των γυναικών. πρόκειται για μια, ένα αντιδραστικό λαϊκιστικό κίνημα που λέει ότι δεν έχει συμπλέγματα, αλλά ούτε εμείς έχουμε συμπλέγματα. να πάμε μπροστά φιλοευρωπαϊστές χωρίς συμπλέγματα.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 Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπνευσμένη ομιλία σας για την Ευρώπη των ανθρώπων, μια ομιλία που δίνει ε, ελπίδα και θάρρος. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τις γυναίκες. Έχουμε διαπραγματευτεί στο Κοινοβούλιο εδώ και πολύ καιρό μια έκθεση που προβλέπει οι άντρες και οι γυναίκες να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στα διευθυντικά συμβούλια επιχειρήσεων. Εσείς ε, μιλήσατε υπέρ της ιδέας αυτής και ε, απευθύνομαι και στον ε, Πρόεδρο Ταγιάννη. Κατά τον χρόνο ομιλίας φροντίζεται εξίσου να μιλούν οι γυναίκες ώστε να μην έχουμε ανισορροπία διότι για να λύσουμε το θέμα της ισότητας θα πρέπει να ακούγεται περισσότερο και η φωνή των γυναικών στο Κοινοβούλιο. Ε, Σα θυμίζω ότι είναι κάποιοι που έχουν υπογράψει την πρόταση τη Κομισιόν. Ε, είμαι ένα από αυτού που έχουν υπογράψει την πρόταση τη Κομισιόν για περισσότερε ε, θέσει για τι γυναίκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το λόγο έχει η κυρία Κοράτσα Μπίλτε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας για την αντιευρωπαϊκή ρητορική από την ακροδεξιά και την ανάγκη για ανανέωση της νομοποίησης ε, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Το Κοινοβούλιο πάντα ψηφίζει ξεπερνώντας τα ε, κομματικά και εθνικά όρια για ενιαία έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε εμείς να αποφασίζουμε που θα συναντιόμαστε και που θα συζητάμε. Και η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Κούρτς μίλησαν υπέρ της μίας έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εσείς ως φιλοευρωπαίος ε, είσαστε διατεθμένοι να στο Συμβούλιο και κατά το προεκλογικό αγώνα να μιλήσετε στους ανθρώπους της Ισπανίας και της Ευρώπης ε, για το θέμα αυτό ή θα αγνοήσετε το θέμα αυτό και θα διακινδυνεύσετε ένα σύμβολο Ευρώπης και συμφιλίωσης στην Ευρώπη, κάτι τόσο αγαπητό σε όλους εμάς, να γίνει ε, σύμβολο σπατάλης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, Revolta Λαντ Μπομφά. Αγαπητέ Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ για την ομιλία που κάνατε. Ευχαριστώ για αυτή την ομιλία που μας δίνει ελπίδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί προτάσει τα κοινωνικά, οικολογικά ε, θέματα, τα θέματα αλληλεγγύης και αξιών και τα ε, θέματα του Ευρωπαϊκού ε, Προϋπολογισμού. Εκφράσατε μεγάλες φιλοδοξίες λέγοντας ότι το 1% του ΑΕΠ των κρατών μελών δεν αρκεί για να έχουμε ισχυρές ευρωπαϊκές προτάσεις. Επίσης, τολμήσατε να μιλήσετε για Ομοσπονδιακή Ευρώπη και αυτό πολύ μας χαροποίησε. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Να επανέλθω στην κατάσταση στην Ανταλουσία. Ανησυχούμε πάρα πολύ εδώ και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να σταματήσουμε κάθε είδους ε, αμφισημία ή παραφύση συμφωνίας ανάμεσα σε, αρχές της σε δυνάμεις της δεξιάς και της ακροδεξιάς. Είναι σημαντικό να τονίζουμε αυτή τη συμμαχία και την ε, προοδευτική αυτή ε, συμμαχία. η τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα διαδικαστικό. Καταρχάς θέλω να απορρίψω και να εκφράσω τη λύπη μου που επιτρέπετε να βάλετε, ε, ε, να, να, να, να αναρτώνται εδώ αφήσει από ε, κρατούμενους. Είναι έλλειψη συμβασμού στον πρόεδρο της κυβέρνησης της Ισπανίας αυτό. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Κύριε Σάντσες. Εσεί ήρθατε ζητώντα να προστατευτεί το ευρωπαϊκό μοντέλο και κάποια άλλα πράγματα από του ακραίου που το απειλούν. Μπορώ να σα πω ότι ε, εσείς μιλάτε για τους ε, εξεμισμούς στην Ευρώπη, αλλά παρακαλώ εξηγήστε μας και σε ολόκληρη την Ευρώπη ότι εσείς είστε πρόεδρος της κυβέρνησης Ισπανίας ακριβώς χάρη σε αυτούς τους εξεμιστές. Δηλαδή, στο του της Καταλωνίας από το χάρη στο του που πάει χέρι-χέρι με τους τρομοκράτες του ΕΤΑ που κατάξει κάποιες φορές ε, ε, έκαναν και πολύ ντροπιαστικά θέματα. Κύριε Σάντσες, πώς μας θα μας εξηγήσετε με, ότι συγκυβερνάτε με αυτού που είναι οι μεγαλύτεροι απαταιώνε τη Ευρωπαϊκή Πολιτική. Ευχαριστώ. Λόπες, Χάβι Λόπες. Πρόεδρε, κύριε ε, φέρατε εδώ τη φωνή των φιλοευρωπαϊστών υπέρ μιας κοινωνικής Ευρώπης που φροντίζει την ε, επισφάλεια των θέσεων εργασίας κλπ. Μια Ευρώπη οικολογική η οποία ηθήνεται του αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Μια ανοιχτή Ευρώπη η οποία θεωρεί ότι η ανοχή και απέναντι στον άλλον είναι λόγος ε, ύπαρξης. Μια Ευρώπη φεμινιστική που θεωρεί την ισότητα των φίλων έμβλημά τη. Αυτή είναι η φωνή της Ισπανίας σήμερα. Μια φωνή που χρειαζόμαστε οι Ευρωπαίοι και που γίνεται καλώς δεκτή από αυτό το σώμα. Μια Ευρώπη η οποία κατανοεί ότι το μέλλον της θα περάσει μέσα από την ε, ε, οικοδόμηση μιας κοινή ε, ηθαγένειας και μετατρέπει τον διάλογο και την συμβίωση σε λόγο ύπαρξή της. Επίσης στην Καταλωνία προσπαθείτε να ξεκινήσετε τον ε, διάλογο ε, ε, επιστρέφοντας πολιτικές λύσεις. Αυτή είναι η μόνη λύση για το μέλλον των Καταλανών, ο διάλογος. Ο κύριος Σωμάτο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Σάντσεθ, ε, περίμενα τουλάχιστον ε, σε μια μιλία που διέρχεται 37 λεπτά να αφιερώσετε 10 δευτερόλεπτα να αναφερθείτε για παράδειγμα στα Κανάρια. Μιλάτε για, τα, για το μέλλον της Ευρώπης αλλά περνάει και από, αυτή την, και από αυτές τις απομακρυσμένες περιφέρειες που χρήζουν στήριξης. Ε, οι Κανάριοι νήσοι ε, έχουν γίνει τουριστικός προορισμός. Ε, Παρ' όλα αυτά θα έπρεπε να είναι κάτι παραπάνω, ένα υπόδειγμα της πολιτικής συνοχής και πολιτικής αλληλεγγύης. Ο κύριος Ταχάνη τόνισε τη σημασία του και είναι αλήθεια. Εμπιστεύομαι ότι ε, θα αποκτήσει και για σας ε, αυτή τη σπουδαιότητα να εκπληρώσετε, να εφαρμόσετε τις ε, συνθήκες, συμφωνίες με τις περιφέρειες αυτές και να τους δείξετε ότι από εδώ, από την καρδιά της Ευρώπης θα έχουν την, υποστήριξη, την πλήρη μας υποστήριξη. Σας ευχαριστώ. Ε, στην κυβέρνησή σας και στον Υπουργό Εξωτερικών σας, Γιουζεφ Μπορέλ, που ήταν πρώην Πρόεδρος ε, αυτού του Κοινοβουλίου. Θέλω να τονίσω από την ομιλία σας ε, τη λέξη φεδεραλισμός. Η ανάγκη να εξακολουθήσουμε να ζητάμε την οικοδόμηση μιας ομοσπονδιακής Ευρώπης που είναι μια ιδέα για την αναδιοργάνωση και της χώρας μας της Ισπανίας που δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά την αναγνώριση της αρμονίας και την δυνατότητα να ζήσουμε με ελευθερία και ειρήνη. Χρειάζεται αυτό για να προστατεύσουμε την Ένωση και τους πολίτες. Ε, αρμονία που τη χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που χρειάζεται να μεταρρυθμιστεί, να μεταρρυθμίσει της Νομισματικής Ένωσης. Ε, χρειάζεται και ο φορολογικός πυλώνας ε, για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια για την ανεργία. Πρέπει να φτιάξουμε μια πλειοψηφία για τις πρόκειτες επόμενες εκλογές με την Κομισιόν ε, για να έχουμε μια ασφάλιση για την ανεργία που να προστατεύει τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ο κύριος Μίγιαν Μόν. Από την ένταξη της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το θέμα της, ε, ε, των σχέσεων της Ισπανίας με τη Λατινική Αμερική ήταν σημαντικό για κάθε Ισπανό ηγέτη. Πώς σήμερα αποφύγατε να αναφέρετε όχι μόνο τη Βενεζουέλα, αλλά και τις πολύ σημαντικές διαπραγματεύσεις με το Μερκοσούρ, κύριε Πρόεδρε, στην ομιλία σας. Μ' αυτό που είπατε, με ανησυχούν αυτό που είπατε, αλλά και αυτά που δεν είπατε. Κάτι ακόμα που θέλω να τονίσω είναι το Brexit και συγκεκριμένα τα θέματα Θα ήθελα να σας ζητήσω στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τον Brexit που θα δούμε πώς θα ολοκληρωθούν να προσέξετε όχι μόνο το Γιβραλτάρ που οπωσδήποτε πρέπει να το προσέξετε αλλά και το θέμα των σαλίας και της αμοιβαία πρόσβασης σε νερά και πόρους. Πολλά συμφέροντα ευρωπαϊκά, ισπανικά και τις περιοχές μου της Γαλλικίας. Ε, ε, θέλω να σας τονίσω ότι το νέο πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο και τα νομικά, νομοθετικά κύματα της Κομισιόν δεν αφήνουν σε καλή θέση τις περιφέρειες της Ισπανίας που μπορεί να υποστούν μεγάλες περικοπές. Παρακαλώ να το προσέξετε πάρα πολύ. Sehr geehrter Herr Präsident, ich freue Κύριε Πρωθυπουργέ, χαίρομαι που μας κάνατε σήμερα την τιμή να βρίσκεστε εδώ σήμερα. Ελπίζουμε σε εσά, ελπίζουμε ότι με το νέο ύφο σας στην πολιτική θα βοηθήσετε να προοδεύσει η Ισπανία. Αντί για αντιπαράθεση, ε, ε, στις ε, διαπραγματεύσεις ε, έχετε εισάγει ένα πιο συνενετικό κλίμα και αντί για πολιτική λιτότητα ε, προσπαθείτε να δημιουργήσετε οικονομικά κίνητρα για οικονομική ανάπτυξη και ισορροπημένο προϋπολογισμό. Ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Όσον αφορά τα μέτρα στην αγορά εργασίας, ε, ανακαλείτε τα μέτρα της, ε, του προκατόχου σας που προσπάθησε να ε, περιορίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχει το λόγο ο κύριος Σάντσεθ για να απαντήσει ερωτήσει των Ευρωβουλευτών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ όλους τους Ευρωβουλευτές που αξιοποίησαν την ευκαιρία γόρευσης. Και θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω γιατί πραγματικά ε, αυτή η ένταση ζω, ζωγονεί την ε, συζήτηση. Υπήρξε μεγάλος αριθμός παρεμβάσεων διαφορετικού πολιτικού στίγματος. Εγώ θα προσπαθήσω να απαντήσω στο σύνολό της, όχι την καθεμία ξεχωριστά βάσει των αξώνων, ε, των θεματολογικών ε, αξώνων τους. Ε, και καταρχήν όσον αφορά τον, το πολυμερές πνεύμα και τα όσα αναφέρθηκαν για τον φεντεραλισμό. Είπα ότι η κυβέρνηση υπερασπίζεται την πολιτική ατζέντα πολιτικής αλλαγής. Πιστεύουμε ε, την ατζέντα 30 βάση του ενός, πολυμερούς, ενός πνεύματος πολυμερούς συνεργασίας. Και θεωρώ ότι συμφωνεί με τα όσα είπα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ισότητα των Φύλων και επίση, τα όσα κάνουμε στην Ισπανία, την έγκριση κάποιων μέτρων που αφορούν την, τον αγώνα κατά τη ε, έμφυλη ε, βία, υπέρ τη ισότητα των φύλων ή την έγκριση νόμων που μειώνουν το μισολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον. Και θα ήθελα εδώ να προσθέσω κάτι. Ορισμένοι παρεμβαίνοντες μίλησαν για την ανεργία που είναι απαράδεκτη στην Ισπανία με σχετικούς ε, χώρους, αν συγκρίνουμε με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όσον αφορά την ένταξη στην Ευρωζώνη. Αλλά επίση θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν... Ε, ε, είναι η πρώτη φορά όπου 48% ε, των όσων είναι κοινωνικά ασφαλισμένοι στην Ισπανία είναι γυναίκες. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ισπανίας που οι γυναίκες έχουν ενταχθεί με τον τρόπο αυτό στην αγορά εργασίας. 22% ε, έχουν ελάχιστες ε, αποδοχές. Είναι πρώτη φορά στην ιστορία, στη δημοκρατική ιστορία της χώρας μας, όπου ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γυναικών είναι καλυμμένοι από το ασφαλιστικό σύστημα. Άρα λοιπόν η ισότητα των φύλων, επίσης αγώνας κατά της ε, παιδικής φτώχεια. Εμείς ε, όχι μόνο θέσαμε την ανάγκη ενίσχυσης ε, της εγγύησης για τα παιδιά, αλλά και, και σε ισπανικό επίπεδο προσπαθούμε να πατάξουμε την παιδική φτώχεια ενισχύοντας όλα τα μέτρα που συνδέονται με την εγγύηση για τα παιδιά ε, προσπαθώντας να την μεταφέρουμε από το νοσιακό στο ισπανικό επίπεδο. Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, ορισμένοι ομιλητές αναφέρθηκαν στο βαθμό δέσμευση της ισπανικής κυβέρνησης σε σχέση με το θέμα αυτό. Πρόκειται να εγκρίνουμε σύντομα ένα νόμο για την κλιματική αλλαγή, μια εθνική στρατηγική για την κλιματική μετάβαση, ε, ε, ούτως ώστε η μετάβαση αυτή να είναι δίκαιη ε, σε εκείνες τις βιομηχανικές ζώνες της Ισπανίας να βρεθούν κάποιες λύσεις εν σχέση με όσων πλήττονται. Επίσης, ορισμένοι εμιλητές ε, αναφέρθηκαν σε ένα ευρύ πακέτο δικαιωμάτων και ελευθεριών ε, που εκπώνησε η συντηρητική κυβέρνηση. Μιλήσατε για τον ε, νόμο Φήμετρο, για όλα όσα έχουν να κάνουν με την εργασιακή μεταρρύθμιση και τα διεργατικά δικαιώματα των εργαζομένων στη χώρα μας. Να σας πω τα εξή, σε σχέση με τον νόμο φήματρο είναι τώρα σε διαδικασία τροποποίηση. Ε, και ελπίζω πω θα μπορέσει να εγκριθεί ε, από τον Φεβρουάριο και μετά. Και όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, να σα πω ότι η κυβέρνησή μα ε, προωθεί το κοινωνικό διάλογο. Σε 7 μόνο μήνε έχουμε εγκρίνει ένα σχέδιο για την απασχόληση των νέων για να μειωθεί σε τρία χρόνια το ποσοστό των ε, νέων ανέργων κατά τρία ποσοστιαίες μονάδες. Επίσης έχουμε φτιάξει ένα σχέδιο αγώνα ε, καταπολέμησης μάλλον της επισφάλειας στην αγορά εργασίας ε, και έχουμε διαπιστώσει ε, και μετατρέψει μάλλον διάφορες μορφές συμβάσεων που ήταν παράνομες στην ουσία σε αορίστου χρόνου ε, συμβάσεις. Στη χώρα μας έχουμε 3, 3 ε, εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες που θα βρουν δουλειά, συμφωνία μεταξύ των συνδικάτων και των εργοδοτών με κάλυψη για τα εργατικά ατυχήματα και ούτω καθεξής. Άρα ε, λοιπόν ε, ε, πλευρη προσπάθεια σε επίπεδο ισπανικό αλλά και σε επίπεδο ευρωπαϊκό και θέλω να κάνω δύο ε, επιπλέον ε, ε, σκέψεις που προέκυψαν σε σχέση με την εξωτερική πολιτική και τη σχέση με τη Βενεζουέλα να σας πω ότι η κυβέρνηση της Ισπανίας αλλά και ως αρχηγός αντιπολίτευσης προηγούμενα δεν αναγνωρίσαμε την νομιμότητα των εκλογών της χώρας αυτής ούτε αναγνωρίσαμε τον ε, Μαδούρο. Ε, η απόδειξη είναι ότι δεν ήμασταν παρόντες όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του. Έχουμε συστηματικά ζητήσει και επανελειμμένα από το καθεστώς του Μαδούρο να ελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούμενους. Ε, χάρη στην καλή διαχείριση του Υπουργού Εξωτερικών καταφέραμε να μπορέσουν κάποιοι κρατούμενοι να έρθουν στην Ισπανία και είχα την ευκαιρία μάλιστα να μιλήσω μαζί τους και σίγουρα η θέση που έχει η κυβέρνηση της Ισπανίας ε, για το θέμα της Βενεζουέλας είναι να προσπαθήσουμε να, να φτιάξουμε μια συμμαχία, ένα, μια ομάδα διευκόλυνσης του διαλόγου που θα αποτελείται από χώρες ευρωπαϊκές αλλά και από χώρες της ομάδας της Λίμα δεν συμμετείχαμε στην απόφαση που πρόθεσε η ομάδα της Λίμα και να σας πω ότι η κυβέρνηση της Ισπανίας δεν έχει την ίδια ιδέα. Προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ομάδα διευκόνησης που ακριβώς αυτό που κάνει είναι να επιτρέψει μια διέλευση με το, μια, ένα διάλογο ε, Επίση, θα πρέπει να μιλήσουμε για τη μεταναστευτική κρίση στη Βενεζουέλα. Ε, να πούμε ότι ε, είναι πολλοί οι Βενεζουαλάνοι που ζητούν άσυλο στη χώρα μας, αλλά επίσης η κρίση της μετανάστευσης ε, στην Λατινική Αμερική, στην Κολομβία, Βραζιλία, Χιλή, με πολλές χώρες που μπόρεσα να συζητήσω αυτούς τους μήνες που είμαι πρόεδρος της κυβέρνησης, να σας πω Ω Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Υπουργό μα αλλά και η κυβέρνησή μα προσπάθησε να, να απελευθερώσει πόρου για να βοηθήσει τι χώρε αυτέ ώστε να διαχειριστούν με λογικό τρόπο την ε, εισρωή προσφύγων που αντιμετωπίζουν και ιδιαίτερα την Κολομβία που ε, ε, την οποία στηρίζουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Για τα Κανάρια νησιά, η κυβέρνησή μας ε, να σας πω ότι σε λίγο περισσότερο από 7 μήνες ξεκίνησε τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος των Καναριών και υπέγραψε όλα τα συμβούλια. Δεν, κάνουμε, δεν φτιάχνουμε υπερπεριφερειακές περιοχές, ε, εμεί στηρίζουμε τα δικαιώματα των, ε, της περιοχής αυτής. Και να πω και κάτι γενικά, τέλος σε σχέση με τις ε, παρεμβάσεις ε, του νεκροσώπων, ε, του ΕΛΚ του Λαϊκού Κόμματος και το θέμα της Καταλωνίας. Το είπα και στην Ισπανία και θέλω να το πω και στους Ισπανούς Ευρωβουλευτές. Να σας πω ότι η μερίσια διάταξη της δεξιάς σημαίνει μάλλον περισσότερο χαρακτηρίζεται από την ακροδεξιά σε δύο θέματα. Πρώτον, το να χρησιμοποιηθεί η Καταλωνία, δηλαδή η συνοχή και η συμβίωση, ως ένα στοιχείο για να κάνετε αντίσταση στην κυβέρνηση της Ισπανίας που θα είναι και θα είναι είναι και θα είναι η σοσιαλιστική κυβέρνηση και τηρεί το Σύνταγμα όσο είμαστε στην αντιπολίτευση και όσο είμαστε στην κυβέρνηση. Και θα ήθελα και το Λαϊκό Κόμμα να κάνει το ίδιο εφόσον είναι στην αντιπολίτευση. Δεύτερον, αν πρέπει να δω για να βρω κάποιο τρόπο διακυβέρνησης που αποσταθεροποιηθεί περιοχέ και χώρε, περισσότερο είναι το, το, το ελβετικό μοντέλο και παρά αυτό το οποίο είδαμε μόλι στην Ανδαλουσία. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε της Κυβέρνησης της Ισπανίας. Σας ευχαριστούμε που απαντήσατε στις ερωτήσεις των βουλευτών. Πιστεύω πως αυτή η συζήτηση ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έγινε πολλή λόγος για την Ισπανία, αλλά και για την Ευρώπη ε, για την πολιτική της Βενεζουέλας για μας είναι κάτι σημαντικό. Εμείς υπερασπίζουμε το δικαιώματα των πολιτών της Βενεζουέλας. Δεν μπορούν να πεθαίνουν από την πείνα σε αυτή τη χώρα που δεν υπάρχει ούτε ελευθερία ούτε δημοκρατία. Ευχαριστώ όλους.